Dear colleagues, may we continue? Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε. Σημείο 5. Τροπολογίες όσον αφορά τις συμβάσεις για διαδικτυακέ ε, και άλλες και του αγαθών Εκθέσει κυρία Χαουτάλα. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω για την δίτη αυτή πρόταση. αδελφή με αυτήν που συζήτησαμε προηγουμένως, πήραμε και συμβάσεις επί ψηφιακού περιεχομένου. Η γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς βάσει του άρθρου 54 του κανονισμού αφορά τις ψηφιακές συμβάσεις για υλικά αγαθά. Τα δύο θέματα βεβαίως, οι δύο φάκελοι, έχουν πολλές ομοιότητες. Οι ομάδες εισηγητών και σκιωδών εισηγητών προσπάθησαν να συνεννοηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο για να αυθυγραμμίσουν τις προσεγγίσεις τους. Κάτι το οποίο όμως δεν ήταν και εύκολο. Θα έλεγα ότι έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, ε, να δούμε τι μπορεί να είναι πραγματικά κοινό συναρτήσει των ομοιοτήτων που έχουν δύο αυτοί φάκελοι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν το είπα προηγουμένω. Το Συμβούλιο έχει προχωρήσει περισσότερο, πολύ περισσότερο στο ψηφιακό περιεχόμενο σε σύγκριση με τα υλικά αγαθά και περιμένουν πλέον την γνωμοδότηση, την έκθεση μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε 172 τροπολογίες επί του σχεδίου για τα υλικά αγαθά. Η έκθεση του κ. Αριμών από την Επιτροπή Ιεστορική Αγορά έχει μια προθεσμία για την κατάθεση λέει, των τροπολογιών, το είχε τον Ιανουάριο. Η ΕΜΚΟ ήδη συντάσσει συμβαστικέ τροπολογίε. Πιστεύω ότι πολλές οι τροπολογίες ήδη είναι, είναι και οι βουλευτές και οι πολιτικές ομάδες είχαν χρόνο να διατυπώσουν απόψει. Η συζήτηση ήταν έντονη και ενδιαφέρουσα. Οπότε θα ήθελα να δούμε το θέμα της εγγύηση, της διαβίου εγγύησης, να το συζητήσουμε περαιτέρω. Στόχος λοιπόν αυτών των τροπολογιών είναι να ακούσουμε τη γνώμη σας επί των σημαντικότερων θεμάτων όσον αφορά τη συγκεκριμένη νομοθεσία και να δούμε ποιων θεμάτων θα προσπαθήσουμε να καταθέσουμε συμβαστικές τροπολογίες μαζί με τον κύριο Αριμό της ΙΜΚΟ που είναι ο εισηγητής, ο σκιώδης εισηγητής. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στις συμβαστικές τροπολογίες. Γενικώ λοιπόν, όσον αφορά τις 172 τροπολογίες, θα τις κατηγορηποιήσω σε βασικές θεμαρικές ενότητες. Εκπέκταση πρώτα απ' όλα του πεδίου εφαρμογή. Στο σχέδιο Λέω ότι χρειαζόμαστε κοινού κανόνε για, για τα ένδικα μέσα, την ένωμη προστασία και στο τομέα αυτών. Όμω χρειαζόμαστε ένα λιγότερο πολύπλοκο πλαίσιο για καταναλωτέ και επιχειρήσει. Συνεπώ, προτείνω τροπολογία που επεκτείνει το πεδίο και στι μη επιγραμμικές, μη διαδικτυακέ πωλήσει και εγγυήσει. Είναι 199 κάθετο 44. Πιστεύω επίσης πολύ ότι χρειάζεται μελέτη επιπτώσεων. Περιμένουμε ακόμη την έκδοση της μελέτης επιπτώσεων, η οποία διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις υπηρεσίες του. Δυστυχώς, φαίνεται ότι το σχέδιο μελέτης επιπτώσεων θα το έχουμε τέλη Σε αυτήν την περίπτωση, αν αυτό ισχύει όντω, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε σημαντική συνεισφορά στο κείμενο, όμως ε, θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε κάποιες από τις τροπολογίες που έχουμε ήδη υποβάλει εν τω μεταξύ. Πολλές από τις τροπολογίες, όντως, αφορούν αυτό, την επέκταση του πεδίου εφαρμογή και την καταρριξη του οδηγίας 1944 Κάτι άλλο στο οποίο επικεντρώνουμε την προσοχή μας είναι το επίπεδο εναρμόνισης. Πέρα από την επέκταση λοιπόν του αντικειμένου, του πεδίου εφαρμογή, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε πραγματικά περί του κατά πόσον θα επιδιώξουμε πλήρη εναρμόνιση ή ελάχιστη εναρμόνιση. Πολλές από τις τροπολογίες θεωρούν ότι η μέγιστη εναρμόνιση δεν θα επιτρέψουν στα κρατημέλη να θεσπίσουν ενδεχομένω αυστηρότερη νομοθεσία. Τώρα, για να προστασία, τα ενδικά μέσα. Κάποιε τροπολογίε προσπαθούν να ενισχύσουν το δικαίωμα επιλογή των καταναλωτών και κάποιοι προσπαθούν να επανεισάγουν τι διαδικασίε επιλογή των ενδίκων μέσων και προσπαθούν να αποσαφηνίσουν την ορολογία που χρησιμοποιεί η πρόταση τη Κομισιόν. Ε, εδώ θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Πώς ε, θα ιεραρχήσουμε τα ένδικα μέσα. Βασικά, ο καταναλωτής πρέπει να έχει την επιλογή. Δεν θα είσαι εδώ πάντως τα της κυκλικής οικονομίας καμία περίπτωση. Εν γέννη, να προκρίνουμε βεβαίως την επισκευή εις βάρος της ε, αντικατάστασης. Ήταν και αυτό ένα δίλημα όσον αφορά τις συμβάσεις ε, επί ψηφιακού περιεχομένου αλλά και υλικών αγαθών. Να υποστηρίξουμε λοιπόν τις ε, επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν βιώσιμα εφορικά προϊόντα που μπορούν να επιδιορθωθούν και όχι τις άλλες. Ως προς το περιεχόμενο τώρα των ε, τροπολογιών, να έρθω τώρα στην διαβίου εγγύηση και εδώ έχουμε μια πολύ έντονη συζήτηση. Δεν κατέθεσα πολλές τροπολογίες. Όταν κατέθεσα όμως το σχέδιο, Είπα ότι θέλω να το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί δηλαδή η διαβίου εγγύηση. Μια απλή πρόταση θα ήταν να ζητήσουμε από τους ε, κατασκευαστές να, παράσουν, να παρέχουν μάλλον εμπορική εγγύηση για συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και αν αυτή η υποσχεθήσα, ας το πούμε έτσι, διάρκεια ζωής δεν ικανοποιείται, τότε να αντικαθιστούν το προϊόν. Αυτό δεν πρέπει να επιβαρύνει όμω υπέρμετρα τους κατασκευαστές ούτε να αποβαίνει βάρος τη ευελιξία. Διότι η διάρκεια ζωή εν τέλει θα καθορίζεται πάντα από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστή θα έχει δικαίωμα να μην αναφέρει όμω διάρκεια ζωή. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίε που αφορούν το θέμα. Πάντω η εγγύηση για, όλη τη διάρκεια ζωή νομίζω είναι μια καλή αρχή. Τώρα κανόνες συμβατότητας και κρυφά ελαττώματα. Και το προηγούμενο και αυτό οδήγησε σε δεκάδες τροπολογίες, κάποιες ασχολούνται με αρκετά με λεπτομέρειες, με επιλογή διατύπωσης, άλλοι όμως τροποποιούν και το αρχικό κείμενο. Για παράδειγμα, πως σημασία πρέπει να αποδοθεί στις προσυμβατικές δηλώσεις και δεσμεύσεις τι περιμένει ο καταναλωτής και πώς θα διατυπώσουμε ότι ένα προϊόν δεν είναι συνδεμένο με πνευματικά δικαιώματα τρίτων μερών, που περιορίζουν δηλαδή τον κατανοητή εν τέλει. Όσον αφορά το θέμα, στο σχέδιο εγώ έχω προσθέσει μια εγγύηση για κρυφά ελαττώματα. Υπάρχει κάτι τέτοιο σε μερικά κρατημέλη και αυτό θα δίνει το δικαίωμα στους καταναλωτές να ζητήσουν αποζημίωση για ελαττώματα τα οποία δεν ήταν ορατά την στιγμή της υπογραφή της σύμβασης. Γι' αυτό πρέπει να το ξαναδούμε στους σκιοδησίγητες. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι απολύτω απαραίτητη αυτή η ρήτρα, κάποιοι λένε ότι είναι περίτη. Κάποιε τροπολογίες λοιπόν αφορούν και αυτό το θέμα. Και τέλο, τελευταία κατηγορία τροπολογιών που έλαβα, ορισμοί γενικέ αρχέ και άλλα ζητήματα. Πολλές από τις τροπολογίες αφορούν την διευκρίνηση των ε, βασικών αρχών που διέπουν αυτήν την οδηγία. Μια ενδιαφέρουσα διευκρίνηση είναι στην τροπολογία 60 που λέει ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να αφορούν και τις συμβάσεις όπου δεν είναι σαφές εάν ο κατανοητής είναι επαγγελματίας ή τελικός απλός ιδιώτης καταναλωτής. Εάν δεν υπερισχύει η επαγγελματική πτυχή, τότε ο καταναλωτής θεωρείται ιδιώτης καταναλωτής. Επίσης, τροπολογία 86 είναι ενδιαφέρουσα. Και πάλι ενδικά μέσα. Ο καταναλωτής ε, πρέπει να είναι σε θέση να προσφύγει και κατά του πολιτή σε επίπεδο χονδρικής. Αυτέ οι τροπολογίε με βρίσκουν σύμφωνοι, αφορούν και το προήμιο ε, εν μέρη. Η προστασία του καταναλωτή πιστεύω ότι είναι προ το συμφέρον όλων, ανεξαρτήτω ε, πολιτικών πεπιθήσεων. Σίγουρα θέλουμε το τελικό κείμενο βεβαίως ε, να αποτελεί καλό συγκερασμό μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εδώ σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε έναν πόλεμο μεταξύ δικαιωμάτων ε, επιχειρήσεων και ιδιωτών, αλλά να καταλήξουμε σε ένα καλό συγκερασμένο κείμενο, όπως προείπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λαμίτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Άουταλα, την εισηγητριά μας, για την παρουσίαση για τα σχόλια και για τις εκτιμήσεις της για τις διάφορες τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησής της. Ως κοιόδης για το ΕΛΚ θα ήθελα να παρουσιάσω σύντομα το πνεύμα των διαφόρων τροπολογιών που κατέθεσα και εγώ ίδια και να απαντήσω επίσης σε τρία κύρια ερωτήματα που αφορούν τις διάφορες θέσεις μας. Καταρχάς για την αντιστοιχεία λύσεων σε σχέση με τα διάφορα πολίσεων. η σχέση μεταξύ επιπέδων αρμόνισης και προστασίας των καταναλωτών και τρίτο θέμα, οι συμπληρωματικές εγγύησεις πέρα δηλαδή της προθεσμίας, της υποχρεωτικής προθεσμίας νόμιμης εγγύησης. Νομίζω ότι θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, αλλά βλέποντας τις τροπολογίες και ακούγοντας την εισηγήτρια, φαίνεται να υπάρχει μια πλειοψηφία για το θέμα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογή. πέραν δηλαδή των συμβάσεων πώληση εξ ή online. για να μην υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές εγγυήσεις ανάλογα με το είδος ε, πωλήσεων που επιλέγει κανείς. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο συμμερίζομαι κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την προσέγγιση που επέλεξε η Κομισιόν για να επιλέξει τα αποτελέσματα που έχουμε. Οπότε δεν θα το τονίσω αυτό. Όμως, να αναφερθώ συγκεκριμένα σε δύο στοιχεία που φαίνονται ότι συνδέονται και που ανέφερε η εισηγήτρια. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει όσο πιο ευρύ εναρμόνιση γίνεται για να είναι αποτελεσματική η οδηγία. Ο κατακριματισμό της εσωτερικής αγοράς ξέρουμε ότι είναι ένα από τα κυριότερα εμπόδια του ενδοκινοτικού εμπορίου. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση κατακαιρματισμού της εσωτερικής αγοράς. Τώρα για τις ελάχιστες, ε, ελάχιστους κανόνες θα πρέπει να εργαστούμε ώστε να υπάρχει βεβαίω το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, αλλά και προοπτικές βεβαίως βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις μας. Οπότε, κάθε λύση η οποία θα βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση δεν θα μπορούσε νομίζω να γίνει αποδεκτή από το ΕΛΚ. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μια υψηλή προστασία καταναλωτών. Εδώ στην Επιτροπή μας τα ξέρουμε αυτά τα θέματα. Και θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά. Οπότε, εξ ονόματος του ΕΛΚ, είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε συζήτηση για επίτευξη ισορροπίας. Όμω βλέπουμε σε κάποιες τροπολογίε που έχουν κατατεθεί να υπάρχουν θέσεις κάπως αντιφατικέ. Οπότε θα πρέπει να τις λύσουμε αυτές τι αντιφάσει. Δηλαδή μπορεί να θέλουμε ας πούμε σε σχέση με την ε, προηγούμενη οδηγία μια ενίσχυση της προστασίας αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να υπάρχει και μια ευελιξία θα πρέπει λοιπόν αυτό κάπως να το συγκεράσουμε και να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε μια πιο ισορροπημένη και πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Στόχος μας είναι το εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης να μην πλήττεται από κανόνες, αλλά αντίθετα να ενισχυθεί. Να καταλήξουμε δύο θέματα που ανέφερε και η κυρία Χάουταλα εγγυήσεις για την διάρκεια ζωής του προϊόντος και τα κρυφά λατώματα. Εγώ δεν νομίζω θα πρέπει να βρούμε μια μέση οδό, μια χρυσή λύση συμβαστική. Και βέβαια θα μας υποβάλει πρόταση συμβαστική η συγγύτρια και θα προσπαθήσουμε μέσω τροπολογιών να προσπαθήσουμε να βρούμε έτσι μια μέση οδό. Θέλουμε βέβαια να πετύχουμε την κατάλληλη προστασία των καταναλωτών. Ξαναλέω το θέμα αυτό μας είναι προσφυλές, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και όχι αντιφατικοί. Αυτά από μένα και αναμένω με χαρά τις συμβαστικές ε, προτάσεις που θα έχουμε από την συγκήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κ. από την ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ είμαι ο εισηγητής ε, στην Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή και Κοινής Αγοράς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επεξεργαστούμε συμβαστικές προτάσεις. Στην Επιτροπή μας έχουμε συζητήσει για αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Η κυρία Γκέπχατ και εγώ διαπληκτιζόμαστε για το ποιο είναι ο καλύτερος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσω αυτά τα οποία είπε η συγγήτρια. Θα σχολιάσω πέντε σημεία και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Το σημαντικότερο ερώτημα εδώ που τίθεται είναι κατά πόσον μπορούμε να, να βελτιώσουμε το επιγραμμικό εμπόριο, το οποίο βασίζεται σε εμπιστοσύνη του καταναλωτή και επίσης ε, και σε εκείνον ο οποίος ξεκινάει αυτή την ε, περιπέτεια. Μπορούμε λοιπόν να προκαλέσουμε εμπιστοσύνη μόνο εφόσον οι κανόνες που θεσπίζονται είναι απλοί και κατανοητοί. Και ένας κανόνας είναι απλός εφόσον ο κατανοητής και ο έμπορος δεν είναι αναγκασμένοι να καταφύγουν σε δικηγόρο για να κατανοήσουν τον κανόνα. Με βάση τον κανόνα υπαριθμών 99 υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις όσον αφορά τις εγγύησεις

και επίσης και όσον αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εγγύησει. Δηλαδή κάθε χώρα έχει κάνει λίγο πολύ αυτό που επιθυμεί και έτσι προέκυψε μια κατάσταση όπου έχουμε πάνω από 30 διαφορετικές νομικές θέσεις στα 28 κράτη-μέλη. Που σημαίνει αν ανοίξω σήμερα ένα κατάστημα online είμαι αναγκασμένος να έρθω σε επαφή με το δικηγόρο μου ο οποίος θα μου πει και θα μου εξηγήσει ποιο είναι το δίκαιο του καταναλωτή σε μια άλλη χώρα. Αυτό οδηγεί λοιπόν στο ότι πολλοί έμποροι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ακολουθούν αυτή την πορεία. Αν όμως θέλουμε ο καταναλωτής να δύναται να έχει προϊόντα από όλα τα κρατημέλη, γιατί υπάρχουν ε, καταστήματα online που πουλάνε σε όλα τα κρατη πρέπει οι κανόνες να είναι σαφείς. Και έρχομαι στην πεμπτουσία του θέματος. Ε, πώς μπορούμε τους κανόνες που θεσπίσαμε παλαιότερα να τους απλουστεύσουμε. Γιατί το 1999 είχαμε μία οδηγία και τότε κάθε κράτος μέλος ε, μπορούσε ε, να προσφέρει στους ε, καταναλωτές και στους εμπόρους περισσότερα δικαιώματα. Η Κομισιόν ακολούθησε μία διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή προσπάθησε να αναρμονίσει συγκεκριμένα δύο-τρία δικαιώματα, έτσι ώστε τα δικαιώματα αυτά να είναι τα ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αν θέλουμε να απλουστεύσουμε τους κανόνες, τότε κατά την άποψή μου όλο αυτό έχει νόημα. Αν θέλουμε έναν καλό κανόνα, τότε θα πρέπει ε, να έχουμε βαθμό εναρμόνισης όσο το δυνατόν υψηλότερο. Άρα δηλαδή και στα 28 κράτη θα πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανόνες. Αυτός είναι ο στόχος. Αν θεωρούμε ότι αυτός δεν είναι σημαντικός ο στόχος και κάθε κράτος μέλος μπορεί να συνεχίσει να κάνει ό,τι θέλει, νομίζω ε, κακώς κάνουμε όλο αυτόν τον κόπο, ε, γιατί όχι να αφήσουμε αυτά που ορίστηκαν το 99 να ισχύουν και σήμερα. Ο στόχος μας είναι η μέγιστη εναρμόνιση. Και όπως σας είπα, διαφωνώ με την κυρία κυρία το πόσο όλα αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε με την προστασία του καταναλωτή. Εγώ πιστεύω πράγματι θα πρέπει να αυξήσουμε την προστασία του καταναλωτή, αλλά το ερώτημα που τείτε είναι κατά πόσον θα πρέπει να πάμε στο ανώτατο υψηλό επίπεδο που υπάρχει σε κράτη-μέλη, αδύνατο αυτό κατά την άποψή μου, ή ε, κατά πόσον γενικά θα πρέπει να αυξήσουμε κάπως την προστασία του καταναλωτή. Όσον αφορά τα ε, ένομα μέσα και την ιεράρχησή τους, ε, συμφωνώ, δεν πρέπει αυτή να καταργηθεί, γιατί σήμερα η τάση είναι και στο Κοινοβούλιο να επικρατεί η κυκλική οικονομία. Αν λοιπόν πράγματι ενστερνιζόμαστε την κυκλική οικονομία, τότε τα πράγματα που αγοράζουμε θα πρέπει να τα επισκευάζουμε όταν παρουσιάζουν ελαττώματα και όχι να τα πετάμε αυτό που θα μπορούσαμε να καταλήξουμε ως ε, συμβαστική πρόταση, δηλαδή καμία εράρχηση και άμεση καταγγελία της σύμβασης και από την άλλη υποχρέωση επισκευής, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι η όλη κατάσταση να είναι πιο απλή. Ε, life span. Αυτή η ιδέα έχει κατατεθεί και σε εμά. Εμείς θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή την ιδέα η ιδέα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και όσον αφορά την κυκλική οικονομία, όμως αν τελικά η ιδέα αυτή πρέπει να μεταφραστεί σε πραγματικότητα, τότε δεν θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν ε, επιπρόσθετο βάρος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά που κάνουμε εδώ δεν ισχύουν ε, για την Amazon, αλλά ισχύει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Ως εκ τούτου να έχουμε κατά νου να μην επαυρύνουμε ιδιαίτερα διοικητικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα κρυφά ελαττώματα, εγώ στη δική μου την έκθεση προτείνω η χώρα η οποία έχει ήδη αυτή την αρχή ε, των κρυφών ελαττωμάτων, εκεί να τα αφήσουμε όσο έχουν τα πράγματα και μετά κάθε χώρα να κάνει αυτό που επιθυμεί. Και πάω στο τελευταίο ερώτημα που είναι αυτό το οποίο παρουσίασε πάρα πολύ ωραία η συνάδελφος Λεγκρίπ, δηλαδή να καταλήξουμε σε μια ισορροπία. Ισορροπία ανάμεσα σε υψηλό βαθμό εναρμόνισης και υψηλό βαθμό προστασίας του καταναλωτή. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε μια ισορροπία. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία με τα οποία μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβασμό. Αυτό θα πρέπει να είναι το πνεύμα που να μας διέπει και να μην λέμε αυτής εξ αρχής όχι δεν γίνεται δεν είναι σωστό. Ε, αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει κοινή αγορά ε, με σαφείς κανόνες, γιατί αν όλοι βάλουν λίγο νερό στο κρασί του, νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω καταρχάς τη φίλη μας, την συγγήτρια, για την πολύ καλή εργασία της, που συνοδεύεται από κάποιες τροπολογίες όπως οι δικές μου. Να πω ότι είμαι υπέρ της επέκτασης του, σχεδίου, του πεδίου εφαρμογή όσον αφορά την πρόταση αυτή ώστε να περιλάβουμε όλες τις μορφές πωλήσεων και αυτές τις διαζώσεις. Και για την περίοδο συμμόρφωσης από δύο χρόνια σε έξι μήνες τόσο και για τις online πωλήσεις όσο και για τα απτά αγαθά. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία νομίζω μεταξύ ασφάλειας δικαίου, ελευθερία συμβάσεων και προστασίας του καταναλωτή. Υπάρχει άλλο ένα θέμα επίσης σημαντικό την κοινοποίηση του δικαιώματος ακύρωση της σύμβασης εκ μέρους του καταναλωτή. Αυτά είχα να πω κυρίω, αλλά να τονίσω επίσης ότι έχω σοβαρές αμφιβολίες για τη θέσπιση διάρκεια ζωής για όλα τα προϊόντα. Επειδή καταρχάς αυτό επικαλύπτεται με την εμπορική εγγύηση που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, έχουμε δηλαδή εδώ μια πόλη ενός ε, πλεονεκτήματος συγκριτικού και έχουμε ένα επιπλέον βάρος, δηλαδή θα πρέπει να καθορίσουμε τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος ανάλογα βέβαια με τις χρήσεις που θα κάνουν, που θα καταναλωτές. Αυτό είναι νομίζω πολύ περιπλοκό. Επίσης, η εφαρμογή αυτού του στοιχείου σε αυτόν τον οργανισμό δεν μου φαίνεται σωστή. Να πω κάτι επίση τελειώνοντα ότι είμαι πεπισμένος ότι θα συνεργαστούμε θαυμάσια με την συγγήτρια και τους σκιώδης ώστε να έχει το σοβαρό και σημαντικό αυτό κείμενο την πλειοψηφία και στήριξη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και Αγκέφχαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πράγματι, κύριε Ρημό, ε, διαφωνούμε με καλοσύνη και αγάπη βέβαια, αλλά Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι η δική μου η πολιτική ομάδα έχει σαφεί απόψει για το τι επιθυμούμε. Ωστόσο, αυτό το είναι απαραίτητο να τσακωνόμαστε. Νομίζω ότι αυτά που προτείνει η κυρία Χάουταλα, δηλαδή το πεδίο εφαρμογής να επεκταθεί σε μη διαδικτυακές πωλήσει, αυτό είναι πολύ λογικό. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχουμε, θα έχουμε διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις για διαδικτυακές και μη διαδικτυακές πωλήσει τη στιγμή που ε, αυτά τα δύο είναι κάπου ρευστά. Στο τέλος δεν ξέρει κανείς τι είναι διαδικτυακό και τι όχι. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη της ε, πολιτικής μου ομάδας. Και εμείς έχουμε καταθέσει και τις ε, σχετικές ε, τροπολογίες. Όσον αφορά το βαθμό εναρμόνισης και τις εγγυήσεις, θα σας πω αυτά τα οποία είπα και προηγουμένως ε, στο ψηφιακό περιεχόμενο, δηλαδή είμαι πρόθυμη να δεχτώ την πλήρη εναρμόνιση αν τελικά είναι υψηλή η προστασία του καταναλωτή. Αν δεν είναι, τότε δεν μπορώ να δεχτώ τα υπόλοιπα. Το ένα είναι συνάρτηση του άλλου. Ως εκ τούτου σήμερα δεν μπορώ να σας πω αν δέχομαι την πλήρη εναρμόνιση ή όχι, γιατί σας λέω αυτό εξαρτάται και από το επίπεδο της προστασίας του καταναλωτή. οχι γιατι σας λεω αυτο εξαρταται και απο το επιπεδο της προστασιας του καταναλωτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αναφέρεται στις, ε, στην εγγύηση των ε, το θέλει ως ελάχιστη εναρμόνιση και αν το δεχτώ αυτό, σε άλλα κράτη όμως οι εγγύησεις είναι μεγαλύτερες. Άρα και τα κράτη θα πρέπει να προσφέρουν λιγότερες εγγύησεις και δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό για τον καταναλωτή. Επίσης αναφερθήκατε σε κάποια ειδικά δικαιώματα ε, αναφέρεστε στη Γαλλία και το Βέλγιο που ισχύουν κάποιες ειδικές διατάξεις, καλά όλα αυτά, αλλά υπάρχουν σε άλλα κράτη διαφορετικές διατάξεις ε, και δεν λύνονται τα προβλήματα. Ας πούμε στο αγγλικό δίκαιο για τις μη διαδικτικές πωλήσει ισχύει το δικαίωμα της ανάκλησης και επιστροφής γιατί δηλαδή να λέμε ε, δεν αλλάζει τίποτα στο Βέλγιο και τη Γαλλία ενώ θα μπορούσε να αλλάξει τη ή κάτι τέτοιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά είναι θέματα επί των οποίων θα πρέπει να εργαστούμε αν πραγματικά επιθυμείτε να υπάρχει ε, πλήρης ε, εναρμόνιση. Και κατά τα άλλα, όσον αφορά την ιεράρχηση των ε, εγγυήσεων, πάλι τίθεται το εξή ερώτημα θέλουμε να προβλέψουμε την ιεράρχηση για όλες τις χώρες και για εκείνες δηλαδή όπου οι πολίτες αποφασίζουν μόνοι τους το τι επιθυμούν. Νομίζω ότι και πάλι εδώ το θέμα της μείωσης ε, της ε, προστασίας του καταναλωτή. Τώρα, όσον αφορά ένα σημαντικό ερώτημα, ε, τη διάρκεια ζωής των προϊόντων να προσφέρεται εγγύηση από τον ε, κατασκευαστή και σας λέω αν δημιουργήσουμε ένα νέο δίκαιο θα πρέπει να δούμε ίσως κατά πόσο θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι στον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε αυτά τα δικαιώματα και παράλληλα με το δικαίωμα της εγγύησης να λέμε και ότι θα προσφέρουμε και μία εγγύηση κατασκευαστή που βέβαια ε, δεν θα είναι ε, πιο περιορισμένη, που θα είναι όμως συνάρτηση της προσδοκόμενης διάρκεια ζωής, την οποία θα ορίζει ο ίδιος ο κατασκευαστής. Δηλαδή δεν λέω ότι αγοράζει κανείς ένα πλυντήριο και έχει διάρκεια ζωής για 20 χρόνια, ο ίδιος ο κατασκευαστής να λέει ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός ε, αντικειμένου. Και αν δεν το θέλει να το κάνει αυτό, αν δεν λέει τίποτα, ο κατασκευαστής έχει αυτό το δικαίωμα Τότε όμως αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στις προκαταρκτικές πληροφορίες του δικαιώματος ε, σύναψης σύμβασης. Αυτό θα ήταν καινοτόμο και θα ήταν και στο πνεύμα της ε, κυκλικής οικονομίας που συζητάμε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε καινοτόμοι, να δούμε λιγάκι ε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό ισχύει και για προϊόντα με βάση την οδηγία Eco-Design για να είναι σαφές ε, ότι πρόκειται για ηλεκτρικά προϊόντα, δεν πρόκειται ας πούμε για ρούχα ή για μολύβια, πρόκειται για προϊόντα ε, για τα οποία μέσω της οδηγίας ε, Eco έχουμε ήδη τοποθετηθεί και πει ότι επιθυμούμε να υπάρχουν βοηθήματα που να διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη, τη μακροχρόνια διάρκεια ζωής των προϊόντων. Έτσι τα έχω φανταστεί εγώ τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπετών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το κείμενο που συζητάμε σήμερα είναι σημαντικό. Οι συμβάσεις πωλήσεων online προλαμβάνουν ένα μεγάλο κύκλο εργασιών για τις επιχειρήσεις και είναι κάτι που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο κατανοητέ. Οπότε πρέπει να ασχοληθούμε. Όλοι συμφωνούμε. Συμφωνούμε επίση ότι θα πρέπει να ασφαλίσουμε την προστασία των καταναλωτών. Όμω, το κείμενο που συζητάμε, κατά την άποψή μου, έχει δύο λατώματα. Το πρώτο, απόβλεψε μία μέγιστη εναρμόνιση, που όπω λέει το ίδιο το όνομά τη, είναι υπερβολική. Να σα υπενθυμίσω ότι η Γαλλική Γερουσία εξέφρασε την ανησυχία τη και θεώρησε ότι αυτή η μέγιστη εναρμόνιση την αρχή της επικουρικότητας. Νομίζω λοιπόν πράγματι έχουν δίκιο, γιατί η συζήτηση που μόλις τώρα κάναμε είναι ένα κείμενο που πάει πολύ μακριά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αυτά που είπε και ο κύριος Καβαντά, ότι θέλοντας να διασφαλίσουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, εδώ μπαίνουμε σε ένα πεδίο πολύ επικίνδυνο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο με τρόπο μειόμορφο να καθορίσουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε διάκριση ανακατηγόρια προϊόντος, τότε συστήνω να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία. Γιατί είναι δύσκολο αυτό. Θα είναι αυτό καταστροφικό. Επίσης, να επιθυμίσω ότι θα πρέπει να δώσουμε δεύτερη σημασία στα βραχεία κυκλώματα και να πω ότι αν θέλετε να το κάνουμε αυτό, τότε θα πρέπει να προωθήσουμε τις εθνικές συμβάσεις πωλήσεων στις χώρες μέλη και να αφήσουμε τις διασυνοριακές συμβάσεις πωλήσεων στο το απαραίτητο. Έχουμε όμω τετραγωνισμό του κύκλου. Δηλαδή θέλω να κάνουμε αυτό αφενός και αφετέρου να έχουμε τις εγγυήσεις. Υπάρχει λοιπόν μια αντίφαση εδώ που θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και δεν βλέπω και κάποιον άλλο να θέλει το λόγο. Κύριε Χάτολα, μήπως θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμα σχόλια. Πέρα από τις τροπολογίες που καταθέσατε ήδη ώστε να διευκρινίσουμε τη βάση εργασία μας για τους επόμενου μήνε. Νομίζω τώρα θα πρέπει να ταιριάξουμε αυτή τη δουλειά με τις θέσεις μας και τις σκέψεις μας. Επειδή νομίζω ότι οι συμβαστικές προτάσεις στην ΙΜΚΟ θα έχουν μεγάλη επίχυση. Ναι, Ευχαριστώ να ακούσω ιδέε για το πώ ακριβώ θα τραγουδήσουμε τον κύκλο, όπω υπόθηκε, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, μεγάλο επίπεδο προστασία καταναλωτών και διασφάλιση το ότι θα έχουμε να κάνουμε με προϊόντα τα οποία θα είναι φιλικά προς τον καταναλωτή, αλλά δεν θα τον παροτρύνουν να υπερκαταναλώνει. Για τις διασυνοριακές πωλήσει Πράγματι θα πρέπει να υπάρχει ένα απλό και κατανοητό πλαίσιο με ασφάλεια δικαίου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και των κατανοητών αλλά και των επιχειρήσεων. Βέβαια ε, υπάρχει το ζήτημα για το πώς θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά τοπικά. Και εγώ βλέπω ότι με τις αγορές online είναι δύσκολο να δει κανεί την προέλευση αυτών των ηλεκτρονικών καταστημάτων, αν βρίσκονται δηλαδή στο Χονγκ στο Λυσίγκη, στο Άμστερνταμ γιατί καλύπτονται με, με μια ώρα έτσι τοπική εικόνα. Είναι δύσκολο. Οπότε θα σας προτείνω σύντομα ημερομηνία για την πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών για να δούμε και τις συμβαστικές προτάσεις που θα υποβάλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο Πρόεδρος για αυτά τα τελευταία λόγια. Πάμε το άρθρο 6 ανταλλαγή με την ΕΟΚΕ σε σχέση με αποφάσεις που έχουν να κάνουν θέματα γάμου κλπ. Γαμικές διαφορές, διαφορές ε, γονικής μέρης κλπ. Ευχαριστώ, κύριε Σβιέσκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που προσκαλέσατε την ΕΟΚΕ. Βλέπω δεν έχετε χρόνο, οπότε θα προσπαθήσω να τα πω γρήγορα. Το σύνθημά μας είναι για την Ευρώπη ενωμένη στη διαφορετικότητα. Εγώ ήμουνα στην ομάδα μελέτης για αυτά τα θέματα δεν είμαι εμπειρογνώμονα. αλλά ο Κριστιαν Μπούρμαν, ο οποίος είναι ο στα συγγνώμη για την απουσία του, αλλά θα προσπαθήσω, μου άρεσε να προσπαθήσω να μεταφέρω τις απόψεις της Επιτροπής μας. Έχουμε εδώ την ελευθερία λοιπόν κίνηση των Ευρωπαίων πολιτών για λόγους εργασίας και άλλους και τώρα έχουμε μικτούς γάμους και παιδιά από αυτούς τους γάμους. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν τη δημογραφική κατάσταση στην Ένωση, αλλά και η νομοθεσία πρέπει να ακολουθήσει αυτό το φαινόμενο. Η ΟΚΕ λοιπόν επιμένει ότι η προτεραιότητα σε περίπτωση απαγωγής θα πρέπει να προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των παιδιών πέραν των εθνικών συνόρων. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να θετηθούν ελάχιστες προδιαγραφές κοινέ για μια διαδικασία κοινή όταν έχουμε να κάνουμε με διεθνή απαγωγή παιδιών. Θα πρέπει να έχουμε κοινέ προδιαγραφέ όσον αφορά την ακρόαση των παιδιών, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά είναι σε θέση να εκφραστούν. Έχουν δικαίωμα να ακουστούν, έστω και αν λοιπόν δεν είναι φυσικά παρόντα, θα πρέπει να υπάρχουν αλλακτικά μέσα, μέσω των οποίων μπορούμε να τα ακούσουμε, α πούμε τηλεδιάσκεψη. Επίσης θα πρέπει να έχουμε επίγοντα προστατευτικά μέτρα που θα επιβάλλονται από τα εθνικά δικαστήρια σε περίπτωση που έχουμε παιδιά προσφύγων που διατρέχουν κίνδυνο. Στις ακροάσεις των παιδιών θα πρέπει επίσης να υπάρχουν άτομα την κατάλληλη κοινωνικοεκπαιδευτική κατάρτιση και συμφωνούμε για το ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα προστασίας των παιδιών. Νομίζω εδώ ότι θα πρέπει να έχουμε ταχείες και αποτελεσματικές ε, λύσεις που να έχουν να κάνουν με τη γονική ευθύνη. Αυτό εξάλλου αναφέρεται και στο άρθρο 55 και νομίζω ότι η αναδιατύπωση αυτού του σημείου είναι ευπρόσδεκτη. Παρ' όλα αυτά στην Επιτροπή μας θεωρούμε ότι η ασαφής διατύπωση αυτού του άρθρου σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μια ασφαλή νομική βάση πάνω στην οποία θα βασιστούν οι χώρες μέλη, οπότε χρειαζόμαστε περισσότερη νομική σαφήνεια. Η Επιτροπή μας καλωσορίζει το γεγονό ότι οι χώρες ε, μέλη είναι υποχρεωμένες να ορίσουν τον αριθμό των ε, δικαστηριών, ανάλογα βέβαια με τα εθνικά δικαστικά, δικαστικά συστήματα. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις της διαδικασίας επιστροφής, και να διασφαλίσουμε ότι οι δικαστές θα είναι σωστά ενημερωμένοι και θα μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με άλλες, ε, με νομικά στήματα άλλων χωρών ώστε να βρεθεί ταχεία λύση. Για τις προθεσμίες των επιστροφών, 18 εβδομάδες, η εντολή επιστροφής θα πρέπει προσωρινά να, εκτελείται γιατί οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει βέβαια αρνητικές επιπτώσεις ε, στο παιδί και στη σχέση του με τους γονείς. Η ΟΚΕ λοιπόν εκφράζει την χαρά τη για τις ευκαιρίες αυτές οι οποίες εντάσσονται περιλαμβάνοντας την πρόταση και θεωρούμε ότι είναι λογικό να υπάρχει μόνο μια έφεση σε σχέση με τι δικασίε επιστροφής. Στις ομάδε μελέτη συστήσαμε κυρίω την ανάθεση των παιδιών σε μονάδες πρόνοιας. Θεωρούμε ότι και επιμένουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι τα παιδιά να πηγαίνουν σε οικογένειε αν αυτό είναι δυνατό. Κατά δεύτερο λόγο, σε αναδόχους και μόνο όταν υπάρχει άλλη λύση, τότε θα πρέπει να μπουν σε δομέ πρόνοια. Έχουμε δύο επιπλέον σχόλια τα οποία δεν αναφέρονται στην έκθεσή μας και είναι τα εξή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να τα καλύψουμε λόγω ακριβώς τη ε, φύση τη μεταβαλλόμενη στι ευρωπαϊκέ κοινωνίε. Καταρχάς, στις περιπτώσεις όπου έχουμε ένα γονέα που δεν κατάγεται από χώρα της Ένωσης. Εκεί συστήνουμε μία διμερή συνεργασία, ιδιαίτερα με τις χώρες αυτές οι οποίες δεν έχουν υπογράψει την ε, συνθήκη της Χάγης για την απαγωγή των παιδιών. Και δεύτερο σημείο, το γεγονός ότι εδώ θα πρέπει να καλύπτουμε τις χαμικές διαφορές Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις γάμου που προσδιορίζονται από εθνικά κριτήρια. Η χάρτα δικαιωμάτων δίνει τη δυνατότητα γάμου. Βέβαια, αναφέρει και την ανέβρεση, τη δυνατότητα ανέβρεση τη οικογένεια και την αφαιρεί χάρτα επίση και την απαγόρευση βεβαίω διακρίσεων ε, για διάφορου λόγου, σεξουαλική ε, προτίμηση κλπ. Οπότε πρέπει να πούμε ότι έχουμε πια στην Ευρώπη νέε μορφέ οικογένεια, νέε μορφέ γάμου και νέε μορφέ χωρισμού. Οπότε αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Ευχαριστώ. Thank you as well. Ε, Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Βεβαίω υπάρχει το θέμα τη επικουρικότητα σε σχέση με αυτό που αναφέρατε στο τέλο τη ομιλία σα. Κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι στο θέμα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τώρα με προστασία καταναλωτών, με εσωτερική αγορά κλπ. Έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά λεπτό και πρέπει να δείξουμε ευαισθησία. Το θέμα είναι και πολύπλοκο, μιλούμε για οικογενειακό δίκαιο. Λοιπόν, όπως είπε ο Πρόεδρος, πρέπει να είμαστε, το λέω για άλλη μια φορά, πολύ προσεκτικοί. Οι αρμοδιότητές μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ συγκεκριμένες. Να δούμε λοιπόν, μάλλον να μην ξεχνούμε, τι μπορούμε πράγματι να κάνουμε εμεί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε τις προτάσεις που ακούσαμε στο Συμβούλιο. Τώρα ο κανονισμό Βρυξέλλες 2 είναι ουσιαστικά τρεις κανονισμοί επί τρία. Τι, τι εννοώ. Έχουμε τις γαμικές διαφορές, έχουμε τη γονική μέρημνα και έχουμε και τα θέματα των διεθνών απαγωγών παιδιών. Και τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, Κρίσιμη θα έλεγα σημασία. για τις ε, οικογένειες, για τη ζωή τους, για το πώς λειτουργούν οι οικογένειες αλλά και τα σύμφωνα συμβίωση και άλλες μορφές συμβίωση. Λοιπόν, η αναδιατύπωση που προτείνει η Κομισιόν του κανονισμού εστιάζεται σε δύο θέματα συγκεκριμένα. Στην εγωνική μέρημνα και στις διεθνείς επαγωγές. Οπότε, ευστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν αναφέρεται στις γαμικές διαφορές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το λέω αυτό και ενώ αυτού που είπε ο εκπρόσωπος της ΕΟΚΕ. Συνεπώς εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε εδώ στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης. Ο μόνος που νομοθετεί όμως, θυμίζω, προκειμένου είναι το Συμβούλιο. Κατά τα άλλα, Είμαστε στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, ότι είναι να εγκριθεί, θα εγκριθεί ομοφόνος. Να ξανά επαναλάβω ότι πρόκειται για πολύ λεπτό θέμα. Επιζητούμε μια συμβαστική λύση, η οποία θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη. Με βάση όλα αυτά έχουμε μια εικόνα του πώς πρέπει να προσεγγίσουμε αυτά τα πολύ λεπτά ζητήματα. Συμφωνώ επίσης ότι η αναδιατύπωση του κανονισμού είναι απαραίτητη. Έχουμε όλο και περισσότερα εντό εωικών διεθνή ζευγάρια, αυτή είναι η ζωή στις μέρες μας. Τα πράγματα συνεχίζουν να αλλάζουν. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των παιδιών στην αυτή κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί δεν πρόκειται πια όπως παλιά μόνο για τα διαζύγια για παράδειγμα. Έχουμε και καταστάσεις όπου δεν έχουμε διαζύγιο αλλά που δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των συζύγων. Και εκεί συμβαίνουν και πολλές απαγωγές, χωρίς να υπάρχει δηλαδή διαζύγιο. Οπότε, αυτά τα προβλήματα έχουμε μπροστά μας, αυτά πρέπει να επιλύσουμε. Έχουμε προτάσεις, τις οποίες θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο, αλλά μην ξεχνούμε ποιος είναι ο υπαρτέτος στόχος. Είναι η βέλτιστη δυνατή προστασία των παιδιών. Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία των γονιών τους. Δεν ανήκουν ούτε σε οργανώσεις, ούτε σε κράτη. Τα παιδιά είναι άνθρωποι. Είναι ανθρώπινες υπάρξεις που χρήζουν προστασίας και σεβασμού. Γιατί τα παιδιά αυτά θα μεγαλώσουν και κάποια στιγμή βεβαίως θα αποφασίσουν για το πώς θα χαράξουν το δικό τους μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι εδώ έχουμε μια τριάδα θεμάτων επί ε, θυμίζω την βράχυνση της διαδικασίας 18 εβδομάδες. 3 επί 6. 3 επί 6 εβδομάδες. Πρώτος βαθμός, δεύτερος και εφαρμογή της απόφασης. Αυτές οι 6 εβδομάδες, οι προθεσμία δηλαδή για κάθε βήμα της διαδικασίας, είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν. Οι 6 εβδομάδες. Όχι παραπάνω όμως. Γιατί? Διότι κάθε καθυστέρηση στη διαδικασία προσφέρει έδαφο στην αξιοποίηση διαφόρων νομικών τεχνασμάτων αμφωτέρωθεν. Και έτσι το παιδί γίνεται μπαλάκι, αν θέλετε, σε ελλείψη νομική, ασφαλείας δικαίου. Όσο πιο βραχή είναι η διαδικασία, τόσο πιο γρήγορα θα έχει κάποιο συγκεκριμένο απότοκο διαδικασία, θα κλείσει η διαδικασία και θα κλείσει και η μάχη για την ε, μέρημνα του παιδιού. Τώρα, για ένα άλλο θέμα, το οποίο έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας καθυστέρησε πάρα πολύ και πολλές φορές ε, για τα μέρη είχε ως αποτέλεσμα σοβαρή οικονομική επιβάρυνση. Λοιπόν, αν θέλουμε να πλουστεύσουμε την κατάσταση για όλους, εγώ είμαι βαθιά πεπισμένος ότι πρέπει να καταργήσουμε την διαδικασία ex equator. Πιστεύω ότι πρέπει οι αποφάσεις να εφαρμόζονται με γνώμονα όμως αποκλειστικά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Εάν δούμε δηλαδή στην πράξη ότι δεν προστατεύεται το συμφέρον του παιδιού, εάν υπάρχει σημαντική μεταβολή στην κατάσταση της οικογένειας, μεταξύ δηλαδή έκδοσης της απόφασης και εφαρμογής της απόφασης τότε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δρομολόγησης διαδικασίας, η οποία θα ανατρέπει, θα κυρώνει την υφισταμένη αποφάση. Κάτι άλλο, όσον αφορά τις διεθνείς επαγωγής παιδιών, πέρα από τις 6 εβδομάδες προθεσμίες που έλεγα λίγο πριν, ένα άλλο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι πώς θα ρυθμίσουμε την ίδια τη φύση της διαδικασίας. Τονίστηκε κατ' επανάληψη, κατά τη διάρκεια ακροάσεων με εμπειρογνώμονες εδώ στην Επιτροπή, το θέμα της ακρόασης του ίδιου του παιδιού. Και εδώ δεν το λέω για να αντιτεθώ ή να αντιταχθώ στις εθνικές διαδικασίες. Ε, βεβαίως, η ακρόαση του παιδιού θα γίνει βάση των κανόνων και των κανονισμών του συγκεκριμένου, του εκάστορε κράτους μέλους. Αυτή η αναγκαιότητα δεν αμφισβητείται. Αυτό αποτελεί και την θεμητοποίηση, την νομιμοποίηση της ε, διαδικασίας. Αυτό τόσο όσον αφορά στην περίπτωση τη γονική μέρημνα, όσο και στις περιπτώσει επαγωγών. Δηλαδή, αν το ένα παιδί είναι σε θέση να διατυπώσει γνώμη, άποψη, προτίμηση, τότε πρέπει όντως να του δοθεί η δυνατότητα να το πράξει. Με τρόπο ουσιαστικό. Αλλά πρέπει να συμβαίνει αυτό, να γίνεται στην πράξη. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανατροπής ακύρωσης της διαδικασίας. Αυτή είναι η προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει. Προς τούτο όμως πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εφαρμόζεται ο κανονισμός. Οι υποθέσεις λοιπόν πρέπει να παραπέμπονται σε δικαστήρια που οι δικαστές ε, έχουν παρόμοια εμπειρία, είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες αποφάσεις και με γνώμονα βεβαίω πάντοτε το συμφέρον του παιδιού. Αυτά τονίζουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τώρα, δικαστική συνεργασία και δικαστική αρρωγή μεταξύ των κρατών μελών. Εδώ δεν ε, μιλούμε μόνο για τα δικαστήρια, αλλά και για οργανώσεις που γνωρίζουν τις ανάγκες των παιδιών, τα δικαιώματά τους, που μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη και μπορούν να παράσχουν τις ε, απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την ε, βέλτιστη ακολουθητέα διαδικασία. Ξέρετε, στο πλαίσιο της συζήτησή μας δεν θα καλύψουμε τα πάντα, ούτε όλα μπορούν να κρυθούν από τα δικαστήρια. Ενώ ότι υπάρχουν και δυνατότητες διαμεσολάβησης εντός της οικογένειας. Να μην το ξεχνούμε. Πολλέ φορέ αυτό μπορεί να είναι πιο εύκολο και προ το συμφέρον του παιδιού. Μια άτυπη διαδικασία με την μεσολάβηση διαιτητή είναι προσφορότερη σε σύγκριση με το αυστηρό περιβάλλον ενός δικαστηρίου. Κάτι το οποίο μπορεί να έχει και επίπτωση βεβαίως στην καλή ψυχολογία των μερών. Οπότε, νομίζω ότι είναι επίσης καλό να ενθαρρύνουμε του, τα μέρη της οικογένειας να προσφεύγουν στη διοίκηση πριν φτάσουν στο δικαστήριο. Θεωρώ ότι δεν θα πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στην εφαρμογή δηλαδή του κανισμού εάν επίσης δεν φροντίσουμε να εκπαιδεύσουμε κατάλληλα όλους τους εμπλεκόμενους στις σχετικές διαδικασίες πάντοτε με γνώμονα του συμφέρον των παιδιών. Ελπίζω ότι Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης, το European Training Network για δικαστές, θα μπορέσει να συνδράμει. Ελπίζω να έχουμε πρόσβαση στο δίκτυο αυτό. Και ελπίζω και ότι το δίκτυο θελήσει να συμμετάσχει και να μας βοηθήσει να, και να διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Ο γνώμονάς μας και φάρος μας είναι πάντοτε τα συμφέροντα των παιδιών. Γι' αυτό συζητούμε εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό κάνουν και τα άλλα θεσμικά όργανα. Προσβλέπω λοιπόν σε περαιτέρω συζήτηση με τους συναδέλφους μου. Γνωρίζω ότι το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, εξαιρετικά λεπτό. Βεβαίως πολύ το έχουν δει πολύ ζεστά, δικαίω. Ευελπιστώ ότι θα πείσουμε όλοι μας, όλοι μαζί, το Συμβούλιο να υιοθετήσει μια πρόταση ισορροπημένη, η οποία θα μπορέσει να γίνει αποδεκτή και από όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, Κυρία Γκέπχαρτ, παρακαλώ, ε, αν έχετε την καλοσύνη, όμως να έχετε και κατά νου ε, το χρόνο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστώ και τον κύριο Σέφκα και την κυρία Σάμα. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπαν και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικά. Εγώ θα εστιάσω την προσοχή μου στην ε, γονική ευθύνη και στην απαγωγή του παιδιού, γιατί νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο θέμα. Κύριε ε, Σεύκα, χαιρετίζω το ότι βεβαίως και θέλετε να βάλετε στο επίκεντρο όλης αυτής της ιστορίας το συμφέρον του παιδιού. Προφανώς και αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης ε, του κανονισμού. Ως ε, πρώην διαμεσολαβήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχω επισκεφτεί πολλά δικαστήρια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το γεγονός ότι μία από τις συστάσεις ε, που είχα συμπεριλάβει στην έκθεσή μου αυτή εμφανίζεται εδώ στο νόμο. Και είναι πολύ ωραίο το ότι ακολουθούνται κάποιες απόψεις. Εδώ αναφέρουμε κυρίως το δικαίωμα του παιδιού στο να εκφράσει την άποψή του. Συμφωνούμε επ' αυτού. Κατόπιν πρόκειται για την συγκέντρωση των διαδικασιών, δηλαδή ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για ποιε διαδικασίε, γιατί κατά κανόνα δεν υπάρχουν πολλέ διαδικασίε. και υπάρχουν οι δικαστέ οι οποίοι στη δικαστική του ζωή έχουν ακολουθήσει μία και μόνο διαδικασία. Εδώ όμω έχουμε να κάνουμε με πολλέ διαδικασίε γιατί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, διαφορετικοί πολιτισμοί, άλλε διαδικασίε, δηλαδή δεν είναι υπεπατημένοι. Και κατά τα άλλα όσον αφορά την ε, χρονική καθυστέρηση όταν επιστρέφονται τα παιδιά, ότι αυτές ε, πρέπει να καταργηθούν, σημαντικό, όπως επίσης και έγκαιρη συμμετοχή της ε, διαμεσολάβησης. Αυτό είναι καθοριστική σημασία, ότι επιτέλους αναγνωρίζουμε και τη διαμεσολάβηση σε αυτή την υπόθεση, γιατί όπως είπε ο κύριος Τσβίφκα, ε, πράγματι ε, μπορούν να επιληθούν εκ των προτέρων πολλά θέματα που δεν χρειάζεται να πάνε στα δικαστήρια. Αλλά οφείλουμε και να μεριμνήσουμε έτσι ώστε η διαμεσολάβηση να μην οδηγήσει στο να παρεμποδίζονται οι δικαστικές διαδικασίες. Επίσης, συνεργασία των ε, κεντρικών υπηρεσιών να ευαισθητοποιούνται αυτές όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ καλό. Αυτό που βεβαίως ε, το βρίσκω λιγάκι προβληματικό είναι το ότι στο άρθρο 7.1 αναφέρεται για πρώτη φορά ότι όταν μετακομίζει ένα παιδί σε μια άλλη χώρα αλλάζει ο τόπος διαμονής του, ε, μπορεί να ανασταλεί η ήδη δρομολογημένη δικαστική διαδικασία. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί κατ' ουσίαν η απαγωγή του παιδιού είναι προγραμματισμένη. Δηλαδή, ένας γονιός θέλει να εντάξει το παιδί σε μια διαφορετική διαδικασία και αυτό είναι προγραμματισμένο. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Στο άρθρο 20 που αναφέρει το δικαίωμα του παιδιού στην έκφραση της άποψής του να σκεφτούμε τουλάχιστον στο σκεπτικό να εισάγουμε και κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για αυτή την ακρόαση, γιατί υπάρχουν χώρες όπου αυτό ήθιστε, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όπου δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία και νομίζω ότι θα ήταν ίσως λογικό να προβλέψουμε κάποια πράγματα. Άρθρο 38 αφορά στα αίτια της μη αναγνώρισης μιας απόφασης. Εκεί αναφέρεται όρος ε, εμπλεκόμενα μέρη. Ίσως θα έπρεπε να ε, ορίζουμε την αυτά τα εμπλεκόμενα μέρη, τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη. Μα ποιος είναι τελικά άμεσα ενδιαφερόμενος. Αυτό νομίζω πρέπει να το ορίσουμε. Κυρία Ρίγνα, και εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς αυτό το θέμα είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο για μας τους ε, ευρωβουλευτές είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε μία και την ίδια κατεύθυνση. Ε, και το θέμα του συμφέροντος του παιδιού ε, μπορούμε να το ε, επαναφέρουμε συνεχώς. Ποτέ δεν είναι αρκετό. Όλοι πρέπει να ασχολούμεθα με το συμφέρον του παιδιού. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για το ότι μας δώσατε μια καταπληκτική γενική εικόνα για μεμονωμένες λεπτομέρειες ε, και για όλα αυτά τα οποία πρέπει να προβάλλουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε καλές λύσεις. Εγώ να προσφέρω μόνο δύο πράγματα. Την κατάργηση αυτής της ε, διαδικασίας. Ε, νομίζω αυτό ε, πράγματι οδηγεί στο να έχουμε δικαιολογημένες επιφυλάξεις σχετικά με την διαδικασία εξακουατόρ. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι σχετικά με την ακρόαση του παιδιού. Βεβαίως και στα διάφορα κράτη υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η διαμεσολάβηση είναι πολύ σημαντική, είναι κάτι για μας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί πιστεύω ότι όπως και εσύ το είπες αυτό προηγουμένως, ντεους, ε, πράγματι έχουμε να κάνουμε μια ειδική περίπτωση. Άρα δηλαδή εδώ θα πρέπει να μπούμε περισσότερο στις λεπτομέρειες. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ε, εορτάσαμε το Ιωβιλέο της Νομικής Ακαδημίας του Τρίρ. Ε, είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να γίνει κάτι και να μην αναφέρουμε έτσι απλά ε, κάποιες επικεφαλίδες, να ορίσουμε ακριβώς ε, πώς σκοπεύουμε να υπηρετήσουμε αυτό το περίφημο συμφέρον του παιδιού. Thank you very much. Uh, Πολύ ωραία, λέει Είχαμε την τελευταία ομιλήτρια για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Και τώρα συνεχίζουμε με το υπαριθμό 17 θέμα που αφορά στο σχέδιο γνώμης για το copyright στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Κάποια στιγμή βέβαια ίσως θα πρέπει να διακόψουμε επ' αυτού του θέματος, γιατί στις 11.30 προβλέπεται να έχουμε ακρόαση. Πες ας ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Thank you, Chair. I understand that we have... Ευχαριστώ πολύ που σημαίνει ότι έχουμε 15 λεπτά για αυτή τη συζήτηση. Εγώ τρία λεπτά θα σας πάρω ε, από αυτό το χρόνο και ξεκινάω με το εξής. Θα ήθελα να σας αναφέρω ε, ποιος είναι ο στόχος μου. Τι είχα κατά νου όταν ε, παρουσίασα αυτό το σχέδιο της έκθεσης. Εγώ αναφέρομαι με γενικούς όρους για τις πιο σημαντικές ε, τροπολογίες τις οποίες κατέθεσα ε, για την πρόταση της Κομισιόν. Όσον αφορά το στόχο, το πλαίσιο, νομίζω πρέπει να έχουμε κατά νου, όπως φαίνεται εξάλλου και από την επικεφαλίδα αυτού του θέματος, ότι μιλάμε για το τα πνευματικά δικαιώματα στην κοινή αγορά, κοινή ψηφιακή αγορά. Ο στόχος λοιπόν είναι ότι αυτά τα δύο μπορούν να συμβαδίσουν. Βεβαίως ε, και πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά πράγματα, ε, στην κοινή αγορά που πρόκειται για την ψηφιακή χρήση και μετατροπή των εργασιών, τη μετατροπή των ψηφιακών διαδικασιών όσον αφορά το text and data, text and data mining. Επίσης να έχουμε κατά νου ότι όλα αυτά θα πρέπει να εξυπηρετούν τον πολίτη. Οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλές προκλήσεις, μερικές εξ αυτών έχουν σχέση με το copyright, τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αλλάζουν συνεχώς οι αγορές και πολλά εξαρτώνται από ένα ε, ιδιαίτερα ρευστό μοντέλο χρήστη ε, υπάρχουν ε, και τέτοιου είδους προβλήματα σε άλλους τομείς ε, όπου επικρατεί η ψηφιακή τεχνολογία, αλλά υπάρχουν και συμπυκνωμένες προκλήσεις, γιατί υπάρχουν και δυσκολίες στην άσκηση των δικαιωμάτων επί των έργων. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε τις σημαντικές προκλήσεις για το copyright σε αυτή την έκθεση. Υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου η ίδια η αγορά έχει προσφέρει και υπάρχουν ε, λύσεις που λειτουργούν. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε αναταραχή σε αυτές τις λύσεις. Όμως οι λύσεις πρέπει να είναι ισορροπημένες, να λαμβάνουν υπόψη όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε κάθε αλυσίδα αξίας. Για να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία του copyright στην κοινή ψηφιακή αγορά χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια, μεγαλύτερη εναρμόνιση, ε, σωστή προσέγγιση των λύσεων που εφαρμόζονται στην αγορά. Για να γίνουν όλα αυτά ε, πρέπει να αποφύγουμε έχουμε την πολλωμένη συζήτηση. Λίγα τώρα θέματα σε σχέση με το περίφημο text and data mining. Ε, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, ε, ίσως διότι οι ορισμοί είναι πολύ περιορισμένοι ή πολύ εκτεταμένοι. Ε, τα ερευνητικά νησιούτα ή μάλλον να το πω εγώ, Αλλιώ, το τι μπορούν να κάνουν τα ερευνητικά Ινστιτούτα, εφόσον το λέμε αυτό, γιατί δεν λέμε και το τι μπορούν να κάνουν όλοι οι άλλοι με τα δεδομένα για αυτό το περίφημο mining. Ε, εγώ λοιπόν ε, θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά και σε άλλου χρήστε τέτοιου είδου δεδομένων. Βεβαίω, αναγνωρίζουμε ότι τα ερευνητικά Ινστιτούτα έχουν προβλήματα, έχουν ε, πρόβλημα να αντιμετωπίσουν αυτέ τι δυσκολίε, Τέτοιου είδου φορέ πολλές φορές σημαίνει ότι ότι πρέπει κανείς να καταβάλει συνδρομή για να υπάρχει μια ευανάγνωστη λύση. Δεν όμως πάντα αυτό απαραίτητο και αυτό ισχύει μόνο σε μια εκδοχή ATDM. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ποιος πληρώνει γιατί. Κατά την άποψή μου, ε, εγώ έχω προτείνει όλα αυτά να τα δεσμεύσουμε με την νόμιμη πρόσβαση. Κατά την άποψή μου, νομότυπη πρόσβαση σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να διαπραγματεύονται μία άδεια με τους εκδότες, εκτός βέβαια αν μιλάμε για πληροφορίες οι οποίες ήδη υπάρχουν και έχουν δημοσιευτεί. Αυτό βέβαια αναπόκειται στις διαπραγματεύσεις. Είτε μιλάμε για μια εταιρεία που είναι startup, είτε μιλάμε για μια φαρμακευτική, εναπόκειται στις διαπραγματεύσεις σε υπονομότυπη εκδοχή να καταλήγουν και σε ε, διαφορετική προσέγγιση. Πάντως ε, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε ήδη ε, την αρχή ότι οι εξαιρέσεις δεν είναι προστίθενται, δεν είναι σωρευτικές. Νομίζω αυτά είχα να σας πω ε, για αυτή τη συζήτηση για το ATDM. Ξέρω ότι η συζήτηση είναι πολύ ευρύτερη, αλλά εγώ πραγματικά προσπάθησα ε, να περιοριστώ. Τώρα, όσον αφορά την διδασκαλία, ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η διδασκαλία και τώρα θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι διαβίου μάθηση. Την εκπαίδευση την έχουμε αφαιρέσει από τα σχολεία και έχουμε εθνικά συστήματα που αναγνωρίζουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ έχω προσθέσει ε, την όχι μόνο των πιστοποιημένων θεσμών αλλά και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πάντως και στη δική μου την πρόταση πρέπει να καταβάλλετε ένα τίμημα αν υπάρχει εμπορικό σκοπό. Το κράτος μέλο. έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιες ε, δημοσιεύσεις ε, ανάλογα με το τι πρόκειται. Μπορούν να αποκλείσουν και ε, σχολικά βιβλία. Αυτά βέβαια θα πρέπει να αφορούν μόνο όσους πράγματι εμπλέκονται στην διδακτική διδασκαλία. Γι' αυτό την διδακτική διδασκαλία ε, και αυτή πρέπει να περιορίζεται χρονικά. Ε, όσον αφορά τα έργα εκτός ε, εμπορίου, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια τροπολογία η οποία κατ' ουσίαν ορίζει και προσαρμόζει αυτά τα έργα τα οποία θα πρέπει να είναι ταυτόσιμα ή και παρεμφερή με τον ορισμό των θεσμών ε, πολιτιστικής εκλειονομιάς που ήδη έχει ρυθμιστεί στην ε, σχετική οδηγία. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, διαφορετικούς κανονισμούς και οδηγίες για το copyright που να περιλαμβάνουν διαφορετικούς ορισμούς για την ίδια ορολογία. Και γι' αυτό έχω αλλάξει την ορολογία. Όμως στις αλλαγές που προτείνω δικαιούχοι έχουν πάντα το δικαίωμα να επιφυλάσσονται αυτοί κατά πόσον θα υπάρχει ε, πρόσβαση στο έργο τους. Εγώ χρησιμοποιώ εδώ τον όρο του να υπάρχουν εκτεταμένες ή ευρείες άδειε και προτείνω και μία τροπολογία όπου δεν υπάρχει διάταξη για αδειοδοτήσεις ή άδειε που να προβλέπουν εξαιρέσεις τότε μπορούμε αυτό να το καθιστούμε, μάλλον να μπορούμε να προσφέρουμε δυνατότητα το περιεχόμενό τους να γίνεται ε, δημοσιοποιήσιμο ακόμα και σε χώρες όπου δεν υπάρχει ευρύ σύστημα αντιοδοτήσεων ή για συγκεκριμένους τομείς οι διαπραγματεύσεις ε, που καθοδηγούνται από κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τα δικαιώματα στη δημοσίευση, άρθρο 11 και τα σχετικά εδάφια, οι ε, εκδότες αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά στην ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση ε, δεν διευκολύνει το περιεχόμενο. Πολλές φορές γίνονται αντιγραφές, αλλά διευκολύνεται η πρόσβαση μέσα από τα συστήματα ε, άλλων μορφών και οι δύο διαδικασίε θα πρέπει να αναγνωρίζονται ω ξεχωριστέ διαδικασίε και δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μία ισορροπημένη προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, εγώ αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να προτείνω μία μέση οδό, άρα προτείνω μία νομική εμπλοκή που σημαίνει ότι προσφέρεται στους εκδότες ε, ένας χώρος ε, στην τράπεζα διαπραγματεύσεων και μία θέση ε, νομικής παράστασης στα δικαστήρια. Το να προχωρήσουμε περαιτέρω, κατά την άποψή μου, σημαίνει ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά και ως εκ τούτου θα είχαμε να κάνουμε με διαφορετικά επιχειρησιακά μοντέλα που σημαίνει ότι ε, έχουμε να κάνουμε με τελείως ε, ρευστά μοντέλα. Το τελευταίο που θέλω να πω για τις ε, πλατφόρμες. Συμφωνώ, χρειαζόμαστε συμβόλαια χρειαζόμαστε τεχνικά μέτρα, αλλά διαφωνώ ότι θα πρέπει να δώσουμε νομικό περίβλημα ε, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και γι' αυτό λοιπόν αναφέρω το παράδειγμα των τεχνικών μέτρων όπως αυτά τα προτείνει η Κομισιόν. Χρειαζόμαστε την προστασία του copyright ε, χωρίς να αλλάξουμε την οδηγία για το εμπόριο ή αν θέλετε προστασία του copyright χωρίς να χάσουμε τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς ε, για τους οποίους αγωνιστήκαμε πάρα πολύ στη σχετική οδηγία. Άρα δηλαδή πρέπει το άρθρο 13 να εφαρμόζεται με ισόρροπο τρόπο και για να το πετύχουμε πρέπει να έχουμε ε, περιορισμένο πλαίσιο, μια σαφήνεια σε ποιον απευθυνόμαστε και ποιο περιεχόμενο μας αφορά. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Before entering into... Ευχαριστώ πολύ. Λόγω έλλειψης χρόνου, να σας πω ότι τα σημεία 9 και 10 θα συζητηθούν στις 4.30 το απόγευμα. 4.30, το 9 και 10 σημείο. Σε λίγο θα αρχίσει και η ακρόασή μας. Και μου ζήσαν το λόγο 7. Είτε λοιπόν θα περιοριστείτε σε ένα λεπτό, είτε Θα ξεκινήσουμε. Μόλις το ζήτησαμε πρώτοι και οι υπόλοιποι θα μιλήσουν στην επόμενη συνάντησή μας και συζήτηση για αυτό το θέμα. Κύριε Ρένταλ. Πρόεδρε, για να είμαστε δίκαιοι, θα ήταν καλό να δώσουμε προτεραιότητα στους σκιώδεις ώστε να μπορέσει να μιλήσει κάθε ομάδα. Ναι, ναι, ωραία. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά αυτό δεν μας λύνει το πρόβλημα του χρόνου. Συγγνώμη, η συζήτηση είναι πολύ σοβαρή και εγώ θα πρότεινα το εξή. Ε, τώρα δεν έχει νόημα να ακούσουμε του και ηγητέ για ένα λεπτό. Αφήστε το, το θέμα να πάει το απόγευμα και να μιλήσουν όλοι. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εγώ αυτό προτείνω. Uh, Ωραία, αποφασίσαμε να κόψουμε κάπως την ακρόαση ώστε να έχουμε 20 λεπτά παραπάνω για τη συζήτηση και μετά ξεκινήσουμε την ακρόαση. Και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Οπότε, Καβαλάης πρώτος Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ την συγκίτρια για αυτή την ε, σοβαρή, στιβαρή δουλειά της. η οποία με έκανε να εκπλαγώ. Η πρόταση τη Κομισιόν μου φαίνεται αρκετά ισορροπημένη και λαμβάνει υπόψη τη τι τεχνολογικέ και ψηφιακέ πρόοδου και προσαρμόζεται στα πνευματικά δικαιώματα. Εδώ λοιπόν έχουμε απόκληση από το αρχικό κείμενο και αυτό θέτει προβλήματα. Υπάρχουν κάποια σημεία που είναι δύσκολο κανείς να υποστηρίξει όσοι έχουν και θα πρέπει πραγματικά να συνεργαστούμε για να πετύχουμε προσεγγίσεις. Έξι σημεία συγκεκριμένα. Το πρώτο αφορά την ευθύνη για τις πλατφόρμες και τον ορισμό τους ως ενεργές πλατφόρμες. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε μια διάκριση με τρόπο ξεκάθαρο τις πλατφόρμες που υπόκεινται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πλατφόρμες οι οποίες υπόκεινται στο κείμενο αυτό εδώ. Άλλο ένα σημείο που θα ήθελα να προσθέσω εδώ είναι ότι οι πλατφόρμες έχουν ένα ενεργό ρόλο στις δημόσιες επικοινωνίες, οπότε θα πρέπει να τις προστατεύσουμε. Δεύτερο σημείο είναι το απαραίτητο και υποχρεωτικό φιλτράρισμα περιεχομένου. Δεν θα πρέπει εδώ να αφισβητούμε τις παρεκκλήσεις για τα πραγματικά δικαιώματα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μέτρα φιλτραρίσματος, τα οποία θα είναι κατά των βασικών ελευθεριών τη στιγμή που η ίδια η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων θεωρεί τα πνευματικά δικαιώματα με τρόπο συγκεκριμένο ως θεμελιώδες δικαίωμα. Οπότε βεβαίως δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αντίφαση. Οι πλατφόρμες είναι αλήθεια ότι φιλτράρουν κάποιο ευαίσθητο περιεχόμενο, δηλαδή περιεχόμενο που, που έχει να κάνει τρομοκρατία, ρατσισμό, αντισημιτισμός, παρακίνηση για μίσος, όλα αυτά λοιπόν για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μηχανισμοί υπάρχουν. Θα πρέπει εδώ να δούμε τι γίνεται τώρα με τους ενδιάμεσους, με τους μεσάζοντες που ήταν μεσάζοντες χθε και σήμερα γίναν πάροχοι περιεχομένου. Οπότε, ας πούμε στην περίπτωση του YouTube, πρέπει να δούμε τι γίνεται με την αναλογία της αξίας η οποία σχετίζεται με τα εισοδήματα, εισοδήματα που έχουν πολιτιστική φύση και που έχουν μια τάξη 66% τεράστιο αυτό. Αυτό όμως βρίσκεται στο περιθώριο της έκθεσης τη στιγμή που μάλιστα το κείμενο της Κομισιόν είναι στη σωστή καθεδρία και είναι προφανές ότι οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν πρόσβαση στην αγορά υπό ίσες συνθήκες ανταγωνισμού. Τέταρτο σημείο αφορά τα γειτονικά δικαιώματα και το άρθρο 11. Νομίζω ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτό ώστε να μην περιορίσουμε την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα σφάλμα στο σχέδιο του κειμένου για τον συντάκτη ο συντάκτης μπορεί πολλές φορές να έχει και ιδιότητα ατόμου που εκπέμπει. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το καθεστώς του. Επίσης, για τα δικαιώματα για την θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται ώστε να υπάρχει σαφήνεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα έντυπο που δεν αποτελείται απαραίτητα από λογοτεχνικά έργα τα οποία προστατεύονται από την οδηγία, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει ας πούμε βίντεο, φωτογραφίες, ε, νέα, νέο υλικό, νέα μορφή ε, υλικό, το οποίο βεβαίω θα πρέπει να προστατεύει και αυτό, να καλύπτεται από τα δικαιώματα γυτνίασης και την επένδυση βεβαίω του συντάκτη, ο οποίο και αυτό θα πρέπει να αποζημιώνεται, αν χρειάζεται. Άλλο ένα σημείο το θέλω να θίξω, το data mining. Συμφωνώ ότι, ότι οι ερευνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να απολαμβάνουν μια εξαίρεση εδώ όσον αφορά τις εταιρικέ σχέσεις οι οποίες έχουν μορφή ΣΔΙΤ. Η έρευνα συνοδεύεται πολύ συχνά από δημόσια κονδύλια, που θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όμως η μέτοχοι σε αυτό το ΣΔΙΤ δεν θα πρέπει να έχουν να κάνουν παρά μόνο με ιδιωτικού φορεί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν δωρεέ ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την έρευνα. Παράδειγμα, η καταπολέμηση του καρκίνου, α πούμε, γνωστό παράδειγμα. Τελευταίο σημείο έκτο, δικαίωμα ισότιμου εισοδήματος για τους δημιουργούς. η δημιουργοί δεν υποβάλλονται σε συλλογικές συμβάσεις. γιατί στις συμβάσεις που έχουν συνάψει περιλαμβάνεται μια κατάλληλη αμοιβή, δίκαιη και αναπαλωτρίωτη. Αυτό αναφέρεται στην αρχική σύμβαση. Και πρέπει να υπάρχει εδώ κάποια μορφή προστασία. Ξαναλέω, πρέπει να συνεργαστούμε για το σύνολο του κειμένου και είμαι στη διάθεση τη εισηγήτρια για να πετύχουμε προσεγγίσεις. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το περιεχόμενο, θα πρέπει να διευκολύνουμε μια πιο ασφαλή πρόσβαση στις πλατφόρμες, θα πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα των δημιουργών και θα πρέπει να βελτιώσουμε τις αμοιβέ τους. Όλα αυτά βέβαια εις όφελος των χρηστών που θα έχουν στη διάθεσή τους διαφοροποιημένο περιεχόμενο ποιότητας και όχι περιεχόμενο που θα είναι ένα είδος fast food δημιουργίας με αντίστοιχους δημιουργούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στραγιάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ διάφανη προσέγγιση σε αυτή την σε αυτή την ε, έκθεση νομίζω ότι αποτελεί συνολικά μια βελτίωση του αρχικού κειμένου της Κομισιόν. Εγώ είμαι ιδιαίτερα υπέρ του να μην δημιουργήσουμε αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία θα περιπλέξουν το σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων. Γιατί ούτω ή άλλω σκοπό τη μεταρρύθμιση αυτή είναι η απλούστευση των κανόνων για, τα, για την ψηφιακή αγορά. Τώρα, για το άρθρο 11 και το τεκμήριο για τους δημιουργούς περιεχομένου. Μπορούμε να συζητήσουμε περιπτώσεις, ας πούμε, όπου συντάκτες μεταφέρουν μη αποκλειστικέ άδειε προς το κοινό. Οπότε γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί, ας πούμε, ο συντάκτης ε, να φέρει περιεχόμενο το οποίο δεν συνοδεύεται από αποκλειστική άδεια. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να προσέχουμε ώστε ας πούμε οι πανεπιστημιακές δημοσιεύσεις θα εξαιρούνται διαφορετικά εδώ ε, θα έχουμε προβλήματα σε σχέση με την ελεύθερη πρόσβαση. Αλλά προσβλέπω βέβαια στη συζήτηση και σε συνεννόηση για να βρούμε μια λύση. Για το 2013 θα πρέπει νομίζω να το ευθυγραμμίσουμε με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ώστε να μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις και περιορισμοί. Παρ' όλα αυτά ανησυχώ με κάποιες προτάσεις του εισηγητή γιατί νομίζω το 17 και το 28 ίσως θα πρέπει να το ξαναδούμε όσον αφορά την ευθύνη. Εγώ ανησυχώ ότι κάπως αυτοί, αυτοί οι όροι, αυτοί οι κανόνες ευθύνης θα πάνε σε τέσσερις οδηγίες και θα είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες. Και το εκτιμώντας 39 αιτιολογική σκέψη 39 νομίζω ότι αναφέρεται σε μέτρα που αφορούν τις πλατφόρμες. Οπότε θα πρέπει εδώ να δούμε και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχουν καθορίσει ξεκάθαρα ότι οι υποπτικές υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίζουμε έστω και εναλλακτικά μέτρα όπως την ταυτότητα ψηφιακού περιεχομένου. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σε κάποιε από αυτέ τι συμφωνίε γενική υποχρέωση υποπτία. Τώρα για το data mining θεωρώ ότι είναι καλή προσέγγιση και συμφωνώ με τι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί σχετικά. Για την εξαίρεση τώρα για την διδασκαλία. για τις άδειε σε σχέση, σε αντίθεση με τις εξαιρέσεις. Είναι δύσκολο τα πανεπιστήμια να βρουν ακριβώς που υπάρχουν άδειε στην αγορά. Και τέλος, η κύρια μου επίκρισε για την ε, έκθεση ότι δεν πάει πολύ πέρα της μη φιλόδοξης πρότασης της Κομισιόν. Εμείς συζητήσαμε την δυσυνολική ανταλλογή και το περιεχόμενο που προέρχεται από χρήστε, κατά το οποίο έχουμε συζητήσει σε διάφορε επιτροπέ και ε, υποεπιτροπέ. Επίση και η διελειτουργικότητα το δημόσιο χαρακτήρα περιεχόμενο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περιλάβουμε εδώ στην έκθεση. Πάντως, ξαναλέω, προσβλέπω στη συζήτησή μα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με την έκθεση αυτή, την οποία αναμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Η κυρία Νίμπλα. Ευχαριστώ πολύ για την ε, έκθεσή σας και θέλω να περιστούμε σε τρεις παρατηρήσεις. Καταρχήν να πω ότι όπως και συνάδελφος κύριος Καβαντά θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι πάρα πολύ ισόρροπη. Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή ε, έχει εξορροπήσει τα πολλά και διαφορετικά συμφέροντα που υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχει ανάγκη συζήτησης και ίσως θα είναι απαραίτητο να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσεις. Από πλευράς αρχής όμως ε, θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι μια καλή πρόταση. Το δεύτερο που θέλω να πω και το ε, θα το πω έτσι συνοπτικά, γιατί αυτό που θα πω αφορά όλες τις ζητήσεις. Κοιτάξτε, η μητέρα των ερωτήσεων είναι η εξής. Θα προστατεύσουμε το έργο του δημιουργού στην Ευρώπη ή όχι. Γιατί αν δεν το προστατεύσουμε, τότε όλες αυτές οι δημιουργικές ε, προτάσεις ε, σε οποιαδήποτε μορφή, είτε είναι κείμενα, είτε είναι ταινίε, είτε είναι βίντεο, οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλου δωρεάν χωρίς ε, στην αλυσίδα της αξίας να υπάρχει κάποια ισορροπία. Κυρίως ε, όσον αφορά την κατανομή των προσποριζόμενων κερδών. Για μένα αυτή είναι η μητέρα όλων των ερωτήσεων και πρέπει να συζητήσουμε από αυτού. Έχω πει επανειλημμένα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή των προσποριζόμενων κερδών και πρέπει να διασφαλίσουμε εκείνη που πραγματικά εργάζονται δημιουργικά στην Ευρώπη, ε, που προκύπτει προς τη θέμενη αξία, αυτοί οι δημιουργοί να έχουν τη δυνατότητα να αμείβονται ικανοποιητικά. Τώρα, στο κείμενο, τρία θέματα θέλω να αναπτύξω. Πρώτον, ε, σχετικά με το text and data mining. Η Κομισιόν ε, πολύ σωστά ε, περιορίζεται σε θέματα έρευνας. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε για λεπτομέρειες, αλλά εγώ είμαι κατηγορηματική. Αυτή την εξαίρεση δεν μπορούμε να την επεκτείνουμε σε όλες τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι εξαιρέσει είναι για εμπορική για μη εμπορική χρήση. Δεν προβλέπονται εξαιρέσει για εμπορική χρήση. Τώρα, άρθρο 11. Η προστασία των ε, δημοσιευμάτων και των ε, τύπου μάλλον. Εδώ τι το ερώτημα. Θέλουμε να έχουμε σοβαρή δημοσιογραφία, ποιοτική δημοσιογραφία. Ξέρετε για μένα την εποχή των fake news είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό είμαι κατηγορηματική ότι δεν μπορούν όλα να είναι δωρεάν, όλα τζάπα, χωρίς να διασφαλίζουμε ότι θα προστατεύουμε κάπως το δημιουργό και όλους τους άλλους που εντάσσονται σε αυτή την αλυσίδα της αξίας. Ε, η πρόταση του άρθρου 11 είναι να ενισχυθούν τα δικαιώματα των εκδοτών. Σωστό αυτό. Ε, υπάρχουν ε, ειδικά δικαιώματα για τους ε, κινηματογραφιστές, ε, για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. άρα δηλαδή σωστό είναι και οι εκδότες να έχουν τα δικά τους δικαιώματα. Και το τελευταίο 13 μεταφορά της λυσίδας αξίας. Εδώ πράγματι πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει καταθέσει μια σωστή πρόταση. Ε, κατανοώ την εισηγήτρια που λέει ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ε, δεν πρέπει να τύγεται. Νομίζω όμως ότι οι προτάσεις που έχουν ε, κατατεθεί αποδυναμώνουν την αρχική πρόταση και εδώ θα ήθελα να επανέλθω στην αρχική διατύπωση της Κομισιόν του άρθρου 13. Ε, χαίρομαι για τις επικείμενες συζητήσεις ε, και θέλω να σας πω ότι εγώ δεν θα επιτρέψω την απεμπόληση της δημιουργικής βιομηχανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να μιλήσω κι εγώ επί του σημαντικού θέματος και του σχεδίου εκθέσεως που συζητούμε. Ανήκω στο ΕΛΚ, στην πολιτική ομάδα του ΕΛΚ, μαζί με άλλους βουλευτές του ΕΛΚ εδώ, που ανέκαθεν υπηρεμήνετο των ε, πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ε, δημιουργών, με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Αυτός είναι ο οδηγός μας. Αυτή είναι η στρατηγική βάση της οποίας θα τοποθετηθούμε επί του θέματος και η οποία θα μας καθοδηγήσει στην συγγραφή των νόμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα σχολιάσω όλα τα θέματα. Θα ήθελα τον χρόνο σας και την προσοχή σας ως προς τα εξής. Άρθρο 11. Συγγενικά δικαιώματα το σχολίασαν συνάδελφοι και ο Ζωμαρή Κεβεντά και η κυρία Νίμπλερ όσον αφορά την, το, το εύστοχο αυτής της ε, διατύπωσης στο άρθρο 11 και τη δημιουργία ακριβώς συγγενικών δικαιωμάτων. Στις μέρες μας η ανεξαρτησία του τύπου απειλείται αν θέλουμε να αναπτυχθεί ο ελεύθερος ανεξάρτητος τύπος, πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερες αμοιβέ, αμοιβή της αξιοποίησης δηλαδή του έργου και της δημιουργίας, της επιγραμμικής δημιουργίας των δημοσιογράφων. Το θέμα λοιπόν αυτό απαιτεί τροποποίηση του άρθρου 11 Πρέπει επίση να ενισχύσουμε το δικαίωμα εκπροσώπηση ενώπιον της δικαιοσύνης. Ίσως να χρειάζεται και συγγενές, συγγενικό δικαίωμα για τα όργανα του τύπου, ώστε να μπορούν να υπεραμείνονται του έργου τους και να εξασφαλίζουν υψηλότερε ε, αμοιβέ. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά, αλλά νομίζω ότι έναντι των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, ε, μόνο η αντίστοιχη κλίμακα μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή προστασία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει εδώ να εξασφαλίσουμε περισσότερη προστασία. Δεύτερον, κατανομή της αξίας καθ' την, το μήκος της αλυσίδας, το value gap, το λεγόμενο στα αγγλικά. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να τροποποιήσουμε και το άρθρο 13 και το εκτιμώντας 38. Νομίζω ότι αυτό εισάγει μάλλον περισσότερη ασάφεια παρά την μειώνει όπως επιδιώκουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να αποσαφηνίσουμε το κείμενο για λόγους ασφαλείας δικαίου. Και το αρχικό κείμενο της Κομισιόν βεβαίως επιδέχεται βελτίωση. Διαφορά λοιπόν με τις τροπολογίες διότι παραλαμβάνω εισάγουν περισσότερη ασάφεια. Διάφοροι οικονομικοί παράγοντες έχουν καταφέρει να παρισφρήσει τόση ασάφεια εδώ που έχουν έτσι ένα, ένα εξαιρετικό εργαλείο για να ξεφεύγουν τις ζωμικές τους υποχρεώσεις. Εδώ θα υποβάλω τροπολογίες για να αποσαφινιστεί το κείμενο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και πιο συγκεκριμένα να πούμε τα πράγματα, ορισμένα πράγματα τουλάχιστον με το όνομά τους. Να πούμε δηλαδή ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους δημιουργούς και την πολισμική πολυμορφία και διαφορετικότητα στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο πλαίσιο το οποίο θα σέβεται τα δικαιώματα όλων των πλευρών. Και για την αμοιβή τώρα των ε, δημιουργών και εκτελεστών, η Κομισιόν και ο εισηγητής νομίζω ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξη επί του θέματος. Ξέρω ότι είναι πολύπλοκο το πρόβλημα, αλλά το θέμα της άμεσης επιστροφής της αμοιβή. Ένα δίρυτο δικαίωμα των δημιουργών να αμείβονται για τη δημιουργία τους, για το έργο τους. Είναι μία από τις πολλές προκλήσεις που βέβαια πρέπει όλοι μαζί να δούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω τους ηγητές. Μετά από τόσες ακροάσεις και συζητήσεις, το αποτέλεσμα νομίζω είναι εντυπωσιακό. Ε, νομίζω ότι δεν έχουμε συζητήσει πολλές, τόσες, ποτέ στο παρελθόν τόσο πολύ μία έκθεση. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για όλο το έργο σας. Λίγα πράγματα τώρα για το σχέδιο έκθεσης. Και εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα για τους εκδότες. Έχουν αρκετά. Ας μην περιπλέξουμε περαιτέρω την κατάσταση. Είναι ήδη αρκετά περίπλοκη από μόνη της. Ας εφαρμόσουμε την νομοθεσία, ας στηρίσουμε τους κανόνες, οι δημιουργοί πρέπει να αμείβονται βάσει του νόμου, δεν χρειάζονται νομίζω νέα και ορφανή δικαιώματα. Όσον αφορά τώρα τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις, ιδιαίτερα για την εκπαίδευση, τη διαβίου εκπαίδευση εκεί, θέλουμε μια εναρμόνιση. Αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να μελετήσουμε την κατάσταση υπέρ των νεοφιών επιχειρήσεων, γιατί αυτές είναι που κρατούν σήμερα την οικονομία. Και το Freedom of Panorama που είπε και το περιεχόμενο παραγόμενο από τους χρήστες. Νομίζω ότι και εδώ χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Είμαι πάντως ε, υπέρ της εναρμόνισης, επαναλαμβάνω, των εξαιρέσεων. Και τέλος, να πω για άλλη μια φορά ότι προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία εκ μέρους των σοσιαλιστών και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας. Πιστεύω ότι θα ήταν το επιστέγασμα μιας ε, σπουδαίας εργασίας Εύχομαι σε όλους μας καλή τύχη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια καλοσυγκυρασμένη έκθεση. Ξέρω ότι έπεσε πολλή δουλειά και από τον εισηγητή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν μακρά η διαβούλευση. Το κείμενο τουλάχιστον αποτυπώνει το περιεχόμενο των συζητήσεων. Πρέπει όμως να διατυπώσουμε ή να επαναδιατυπώσουμε κάποιες βασικές αρχές. Το σημείο κίνησης όλων αυτών είναι πώς βλέπουμε τις αρχές που προσπαθούμε να ενσωματώσουμε στο κείμενο. Για παράδειγμα, ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά που ισχύουν για τον ψηφιακό κόσμο σε όλα τα άλλα. Στη δημοσιογραφία, στις τέχνε, όπου δημιουργείται περιεχόμενο τέλο πάντων και όπου υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αμείβονται αξιοπρεπώς και αυτό δεν ισχύει παντού. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Και για όλους αυτούς που παράγουν περιεχόμενο, που είναι η παραγωγή αν θέλετε, αλλά και πλατφόρμες μέσω που είναι το, το μέσο. Ε, αυτοί είναι βεβαιω υπεύθυνοι, ο νόμος ισχύει και για αυτούς, έχουν και δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως ε, άλλωστε οι εφημερίδες, ε, οι σκηνοθέτες ε, κινηματογραφικών ταινιών, όλοι όσοι εμπλέκονται στην, στον οπτικο-ακουστικό χώρο. Ό,τι λοιπόν ισχύει για τους άλλους, να ισχύει και για τον ψηφιακό κόσμο, όσον αφορά τις βασικές αυτές αρχές. Το επιγραμμικό με το μη επιγραμμικό λοιπόν πρέπει να εξομοιωθούν. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί, αν θέλετε, όσον αφορά τις πλατφόρμες. Εδώ μιλούμε για ενεργητικές και παθητικές πλατφόρμες, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει στην πράξη τέτοια διάκριση. Όλα είναι ενεργά. Ο τρόπος με τον οποίο ανεβάζουν περιεχόμενο οι πλατφόρμες είναι στην κρίση του καθενός. Αλλά κάθε φορά που μπαίνετε, ανεβαίνετε βλέπετε μια πλατφόρμα, είναι στο χέρι σας να αξιολογήσετε το περιεχόμενο, αλλά το κοινό είναι ότι έχουμε μια αποθήκη περιεχομένου, που δεν είναι όμως ποτέ απόλυτο στατικό. Γι' αυτό και οποιαδήποτε πλατφόρμα είναι ενεργητική, διότι θέτει στη διάθεση του κοινού περιεχόμενο και αυτό συνεπάγεται υποχρεώσεις και ευθύνη που δεν έχουμε καταγράψει επαρκώ, νομίζω στο κείμενο. Συνεπώ να είμαστε απολύτως σαφεί. πώς θα χειριστούμε τις πλατφόρμες ε, και βεβαίω εν τέλει να ε, δεσμεύονται οι πλατφόρμες από την νομοθεσία. Δωρεάν ίντερνετ δεν υπάρχει. Όλοι όσοι εμπλέκονται στο διαδίκτυο, όσοι ανεβάζουν περιεχόμενο, εργά, τέχνης κλπ. στο δημόσιο χώρο, φέρουν ευθύνη και πρέπει να υπόκεινται λοιπόν στον νόμο. Και αυτό είναι μια βασική αρχή. Και μια άλλη βασική αρχή είναι ότι όσοι εργάζονται στους σχετικού τομείς πρέπει να μείβονται αξιοπρεπώ. Οι δημιουργοί πρέπει να απολάβουν των απαραγράπτων δικαιωμάτων τους, όπως οι δημοσιογράφοι και άλλοι. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τρομακτικά φαινόμενα όπως τα πλαστές ειδήσει είναι κανόνες. Είναι νομοθεσία για να μην ε, γινόμαστε μάρτυρες καταχρήσεων σε καθημερινή βάση. Γιατί αυτά βλέπουμε συνεχώς γύρω μας. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτά, αλλά πρέπει το διαδίκτυο να το αντιμετωπίσουμε όπως και τον υπόλοιπο κόσμο, τον πραγματικό κόσμο. Νομίζω ότι σιγά σιγά αποσαφηνίζεται πάντως η κατάσταση. Ε, κάπως έτσι βλέπουμε τα πράγματα. Και νομίζω ότι σωστά έπραξε η Κομισιόν. Καλή είναι η προσέγγιση της και η έκθεση είναι καλή. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ, επειδή ξέρω ότι θα ξεκινήσει λίγο η ακρόαση, προσβλέπω σε περαιτέρω συζήτηση. Εγώ με δίστανται ακόμη. Πολύ, πολύ σημαντική η έκθεση. Θα συμμετάσχουμε όλοι στην συζήτηση και ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Ροσχέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Περιμένουμε πολλά από αυτήν την έκθεση, από την πρόταση μάλλον. Ιδιαίτερα δεδομένες της διαπίστωσης ότι ένα μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των έργων της Διανίας ε, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Περιμένουμε αυτή την πρόταση για να επικρατήσει κάποια ισορροπία, να βάλουμε μια τάξη και να δώσουμε στους πνευματικούς ε, δημιουργούς τα μέσα ε, ώστε να συνεχίσουν κανονικά τη δραστηριότητά τους. Η πρόταση της Κομισιόν ήταν ενδιαφέρουσα για τρεις λόγους. Τα υπόθηκαν και προηγουμένως ανάδειξη των εκδοτών του τύπου με τα συγγενικά δικαιώματα, οι πλατφόρμες, το value gap, η κατανομή της αξίας και βεβαίως εν τέλει οι διατάξεις για την καλύτερη αμοιβή και την διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ε, δημιουργών και χρηστών. Έγινε πολύ καλή δουλειά. Το σχέδιο όμω ε, του κειμένου απομακρύνεται από τον αρχικό στόχο. Παρά πολλές καλές προτάσεις παρά την διάρκεια και το βάθος του, διαλέγου, του διαλόγου. Φοβάμαι ότι έχουμε χάσει λίγο το στόχο από μπροστά μας. Το δεδομένο είναι τι κάνουμε γενικώ για το πολιτισμικό μας προϊόν και πώς θα αμείβουμε τους δημιουργούς. Όσον αφορά την διαφάνεια και την αμοιβή των δημιουργών, το κείμενο είναι μάλλον καλύτερο, βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχω στο μυαλό μου κυρίως τα άρθρα 15 και 16 όπως είπα, προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως εξεπλάγει με κάτι άλλο. Εμείς ε, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στον ρόλο του τύπου, του ποιοτικού τύπου στη δημόσια διαβούλευση, στην ενημέρωση, στην ανεξάρτητη ενημέρωση κλπ. Ο ποιοτικό τύπος πρέπει να μπορεί να επιβιώνει χωρίς ε, κόλπα, ούτως υπήν, Λοιπόν, τα συγκεκριτικά δικαιώματα για τους εκδότες είναι μια καλή ιδέα προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί βοηθούν ουσιαστικά στην διάδοση του προϊόντος και αυτοί διαπραγματεύονται και με τον ψηφιακό κόσμο σε μεγάλη κλίμακα. Πολλές φορές και αυτοί γίνονται θύματα καταχρήσεων και πολλές φορές οι αμοιβέ τους καθορίζονται ετεροβαρός. Συνεπώς, Ας πατήσουμε πάνω σε αυτό για να τους προστατεύσουμε καλύτερα. Κάποιοι λένε ότι αυτό οδηγεί σε έλλειψη ασφαλείας δικαίου, αλλά να το δούμε αυτό, γιατί φοβούμαι ότι αν το αφήσουμε το πράγμα έτσι, θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη ασάφεια. Ίσα ίσα. Εγώ θέλω να καθορίσουμε το ποιο κάνει τι και ε, νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε ανυπεράσπιση στους τους εκδότες. Τώρα για τις πλατφόρμες και το λεγόμενο value gap, το χάσμα αξίας, την κατανομή της αξίας στην αλυσίδα. Σήμερα οι πλατφόρμες είναι ενδιάμεση οι οποίοι αξιολογούν το τι θα ανεβάσουν, κοιτάζουν τις διαφημίσεις, το εισόδημα από τις διαφημίσεις που προσδοκούν, φιλτράρουν όπως και να το κάνουμε το περιεχόμενο όχι αναγκαστικά ε, βάσει της αξίας του περιεχόμενου, το θέμα είναι τα, τα έσοδα εν τέλει. Και νομίζω ότι αγνοούν ε, τα πνευματικά δικαιώματα, ε, είτε αυτό αφορά έναν πίνακα, μια φωτογραφία κλπ. Οι πλατφόρμες επίσης είναι υπεύθυνε, φέρουν ευθύνη ότι ανεβάζουν για το αν προστατεύουν τους ανηλίκους για παράδειγμα Μιλάμε για πλατφόρμες με τεράστια κέρδη, τεράστια κέρδη σε σύγκριση με τους πραγματικούς δημιουργούς. Αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι αδίκο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω προς αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή και τις αμοιβέ των δημιουργών. Και για τις εξαιρέσει, τέλος, και αυτό το συζήτησαμε εκτενώς, ε, μια εξαίρεση πάντως κάθε εξαίρεση φοβούμαι ότι είναι απαλωτρίωση των δικαιωμάτων των δημιουργών. Περί αυτού πρόκειται. Στερούμε τον δημιουργό από ένα δικαίωμα. Λοιπόν, όχι. Οι δημιουργοί πρέπει να αμείβονται. Από τη στιγμή που κάποιος ε, έχει μια οικονομική δραστηριότητα πρέπει να πληρώνει. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που για λόγους δημοσίου συμφέροντος το δημόσιο θέλει να διευκολύνει την πρόσβαση και, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αμείβονται οι δημιουργοί. Ίσως με διαφορετικό τρόπο, ε, αλλά και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αμείβονται. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ολοκληρώσουμε προς το παρόν τουλάχιστον αυτή τη συζήτηση και θα τη συνεχίσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Και ευθύς αμέσως ε, ξεκινάμε με την ακρόαση για τις νέες υποχρεωτικές ε, εξαιρέσεις. Κάποια στιγμή, από κάποια στιγμή και μετά δεν θα έχουμε διερμηνία αυτό αν δεν κατορθώσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγμα που μας δόθηκε σήμερα το πρωί. Πρώτος ομιλητής, ε, Αλαβάν Στράβελ, καθηγητής ε, στη Λουβέν, ε, Καθολικό Πανεπιστήμιο και σε άλλα πανεπιστήμια θα μας μιλήσει για τις ακαδημαϊκές προοπτικές το πολύ 6 λεπτά έχετε το λόγο. Το πολύ για 6 λεπτά. Ε, να συστηθώ Είμαι καθηγητής, ε, διδάσκω δίκαιο ε, περί copyright ε, μεταξύ άλλων. Είμαι δικηγόρος, έχω δουλέψει για εκδότες και για εταιρείε πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπώ κανέναν. Μιλώντας εξ ονόματος κάποιου, είναι εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα copyright. Δεν μου έχουν αναθέσει να ομιλήσω εξ ονοματός των σήμερα, αλλά νομίζω ότι δεν θα διαφωνούσαν με αυτά που είπα. Πρόεδρος, αν έχει την καλοσύνη να απομακρυνθείτε από την αίθουσα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας είπα, είμαι κυρίως καθηγητής, που σημαίνει ότι ίσως είμαι λιγάκι σχολαστικός. Είδα την πρόταση της Επιτροπής και η δική μου ομιλία βασίζεται στο κείμενο της Επιτροπής. Δεν μπόρεσα να δω τις ε, ε, τροπολογίες, αλλά πιστεύω ότι ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Πάντως στο κείμενο της Επιτροπής ε, υπάρχουν διαφορετικοί δικαιούχοι και για το text and data mining είναι η ερευνητικοί φορείς. Εγώ δεν έχω ε, κανένα πρόβλημα με το καινούριο κείμενο και θα σας εξηγήσω. Τρεις εξαιρέσεις. Η πρώτη στο κείμενο της ε, Κομισιόν αφορά τα περισσότερα θέματα. Και νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό στο μέλλον να μπορεί κανείς ε, να εξάγει, να επεξεργάζεται δεδομένα. Αυτή είναι μια σημαντική διαδικασία. Και επίσης ε, πρέπει να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ακατέργαστα δεδομένα αυτά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή το copyright ε, κατ' ουσίαν δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά. Ίσως να προκύπτουν κάποια θέματα όταν γίνεται μεταφορά πετρελαίου. Μπορεί να προκύψει υπερχείληση, ζημιές, αλλά δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ε, λοιπόν, πάμε τώρα στον ορισμό του TDM, Text and Data Mining. Υπάρχει ένα στάνταρτ ε, ορισμός που νομίζω συμπίπτει με αυτόν που έχουμε στο σχέδιο της οδηγίας και ε, ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για την απόκτηση δεδομένων, όπως σας είπα προηγουμένως, ε, κατά πόσον υπάρχει θέμα με το copyright, δεν είμαι σίγουρος, γιατί αυτά τα δεδομένα δεν προστατεύονται. Και βεβαίως ο στόχος είναι να υπάρξει ανάλυση, να προκύψουν επιπρόσθετες πληροφορίες, αυτός, αυτό είναι, σημαίνει σωστός ορισμός. Τώρα, τα text and data mining θα πρέπει να καλύπτουν το copyright. Όχι, είναι απάντησή μου για διάφορους λόγους. Κυρίως διότι το copyright βασίζεται στο διαχωρισμό ανάμεσα στην έκφραση και την, ε, που προστατεύεται και την ενημέρωση που δεν προστατεύεται. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με δεδομένα. Αυτό είναι εκτός του πεδίου εφαρμογή του copyright. Νομίζω ότι το TDM ε, δεν έχει άμεση επιρροή στις προστατευόμενες ε, διαδικασίες. Πάντως όπως λέει ο του TDM, δεν επιλέγει κανείς ε, να κάνει μια δουλειά επειδή του αρέσει, απλά προσπαθεί να βρει κάποιους ε, συσχετισμούς ε, και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα αυτά δεν καλύπτονται από το copyright. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι τελικά Εάν το TDM προστατεύεται από το copyright, νομίζω ότι αυτό αντιβαίνει στο στόχο του copyright που είναι να διαδίδει πληροφορίες και γνώση και εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο δεν είναι μόνο δική μου άποψη αυτή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copyright. Το πρόβλημα προέρχεται από το δικαίωμα αναπαραγωγής, ε, άρθρο 2 14 νομίζω έχετε μπροστά σας τον ορισμό όπου όταν γίνεται λόγος για αγορά ε, μπορεί να περιλαμβάνονται και προσωρινά αντίγραφα. Αυτό ερμηνεύτηκε πολύ με μεγάλη ευρύτητα πνεύματος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα γιατί προκύπτουν τα θέματα έχουμε προβλήματα με τα αντίγραφα του TDM αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα αντίγραφα που υπάρχουν στο ίντερνετ και αυτά είναι απαραίτητα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, όλα αυτά τα αντίγραφα κατ' ουσίαν καλύπτονται από την ευρεία ερμηνεία της αναπαραγωγής του ορισμού της αναπαραγωγής. Πρόβλημα υπάρχει με την αναπαραγωγή κάποιων καθαρά τεχνικών αντιγράφων και νομίζω ότι αυτό περιλαμβάνει και τα αντίγραφα του TDM. Αυτή είναι μία ακραία άποψη Βεβαίω, αν εσεί πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα αναπαραγωγή που να καλύπτει τη δραστηριότητα του TDM, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και απαραίτητε εξαιρέσει. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε στο κείμενο της Κομισιόν. Προβλέπονται δικαιούχοι, Αυτή είναι οι ερευνητικοί φορείς. Πόσο χρόνο έχω ακόμα. Έχετε ήδη ξεπεράσει το χρόνο σας κατά 33 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, όπως σας είπα, όλα αυτά καλύπτονται με μια νέα τροπολογία, την 31, που ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Ε, άτομα δεν καλύπτονται από αυτόν τον ορισμό ε, και επίσης και έρευνες που γίνονται από πανεπιστήμια, ούτε και αυτές καλύπτονται και από άλλους ιδιωτικούς φορείς. Ε, σας είπα, δεν καλύπτονται όλα αυτά κάτω από το ε, ερευνητική φορείς ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση, αλλά κατά τα άλλα θα πρέπει ε, να υπάρχει νομότυπη πρόσβαση. Αυτό θα πρέπει να είναι προϋπόθεση στο κείμενο της Κομισιόν. Αναφέρομαι κυρίως στην τροπολογία υπερθμών 31 ε, και δεν υπάρχει και ορισμός του στόχου Στόχο της ε, ερευνητική διαδικασία που λέει Κομισιόν θα πρέπει να υπάρχει και ε, έρευνα για το TDM. Είναι σημαντικό να προσθεθεί αυτό. Κατά τα άλλα ε, δεν είναι πολύ σημαντικά τα υπόλοιπα σχόλια. Ανέφερε και ένα, είδατε ένα αξίωμα που μπορεί κανείς να ακολουθήσει. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να ε, θεωρούμε ότι εδώ πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Τα αυτά που είπα τώρα στο τέλος δεν έχουν σχέση με το copyright. Ευχαριστώ. Ε, thank you, ε, professor. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για την κατανόηση που δείξατε στο χρονικό περιορισμό. Μαρία Ελίζαμπεθ Ρέμπιντερ. Νομικό Συμβουλό στα πανεπιστήμια που ασχολούνται με θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και μέλο μια οργάνωση που ασχολείται με αυτά τα θέματα αυτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ ερευνητικού οργανισμού και βιβλιοθήκε. Μα εικονοποιεί το σχέδιο τη έκθεση χαιρετίζουμε το κείμενο και την αναφορά του στο Text and Data Mining. Ας δούμε λοιπόν από πού ξεκινήσαμε. Ξεκινάμε από τη συνθήκη της Λισαβόνας που αναφέρει ότι η έρευνα δεν αφορά μόνο τα πανεπιστήμια αλλά την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Το αναφέρουμε και εδώ, οπότε ευχαριστώ τον συντάκτη της έκθεσής σας που πήγε στο κατεύθυνση όπως και ο καθηγητής προηγουμένως. Για το άρθρο 2. Βλέπετε έχουμε τους ορισμούς όπου λείπει ο ορισμός του ατόμου ασχολούμαι από το 1994 με τα πνευματικά δικαιώματα και η οικογένειά μου ασχολείται με τα πνευματικά δικαιώματα εδώ και 100 χρόνια. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νομοθετική πράξη, αλλά συνεχίζει να λείπει ο ορισμός του ατόμου. Τα πρόσωπα δηλαδή, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, εντάξει, σωστά όλα αυτά, αλλά ξαναλέω θα πρέπει να προσθέσουμε ένα ορισμό πέραν των φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων. Στο άρθρο 2. Μετά, όπως είπε και ο καθηγητής, δεν υπάρχει προστασία για τα δεδομένα και τις πληροφορίες. Έχουμε μόνο κοινέ μορφές προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, όπως τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τα διπλώματα συγγνώμη και έχουμε κάποια γενικά και όριστα δικαιώματα για τις βάσεις δεδομένων. Οπότε αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, έχουμε πολύ συγκεκριμένα και λεπτομερώς προσδεμένα δικαιώματα στις βάσεις δεδομένων. Γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως νομική προστασία για την πληροφορία και για τη γνώση η γνώση είναι ελεύθερη και η πληροφορία. Οπότε θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι το σύνολο της Ένωσης δεν θα υποχρεωθεί μόνο να ασχολείται με τους συντάκτες, είναι τους δημιουργούς περιεχομένου που έχουν κάποιο πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Θα πρέπει λοιπόν στο άρθρο να το προσθέσουμε αυτό. Με του προσώπου που λέγαμε προηγουμένω, φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσθέσουμε και τα δικαιώματα, τα νόμιμα δικαιώματα που έχουν αυτά τα πρόσωπα, είτε νομικά είτε φυσικά, πανεπιστήμια κτλ. σε σχέση με το data mining. Ξαναλέω λοιπόν, αυτά που γράφετε είναι σωστά, αλλά θα πρέπει στα εκτιμώντα, στα εκλογικέ σκέψει ή κάπου στο διατακτικό να καλύψουμε αυτό το κενό τη έλλειψη δηλαδή προστασία όσον αφορά τα δεδομένα και την πληροφορία. Επίσης, να προσθέσω ότι μπορεί να υπάρχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ οργανώσεων και οργανισμών ερευνητικών και εκδοτών. Αυτά είχα περίπου να σας πω. Έχουμε μία εκδήλωση για τη startup στο Ελσίνκι, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και πρέπει να σας πω ότι σας χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ επειδή μας βοηθάτε όλες τις startups, τις νεόφυτες επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάρλο Ραβιτσάρη, νομικό σύμβουλο στην Διεθνή Οργάνωση Εκδοτών Επιστημονικού και Τεχνολογικού Περιεχομένου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πάω λίγο πίσω στη διαφάνειά μου. Συμφωνώ με την προάλληλη σας και τον καθηγητή και εγώ είμαι καθηγητής δικαίου πνευματικών δικαιωμάτων και σήμερα εδώ εκπροσωπώ εκδότες ιατρικού, τεχνολογικού, επιστημονικού περιεχομένου. το οποίο αφορά το 16 της έρευνας και δημοσίευσεων παγκοσμίω. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα που συζητάμε και εσείς χαράζετε το δρόμο που θα ακολουθήσει η Ευρώπη εδώ. Το text data mining είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό επειδή υπάρχει πληθώρα πληροφοριών. Ήδη πολλές βιομηχανίες όπως οι θερμοκόβιομηχανίες δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτό το data mining. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με την προλαλή σας. Το μέλλον βασίζεται ακριβώς σε αυτό το data mining, το οποίο πρέπει να λαμβάνει η χώρα πριν πάμε στη μορφή, μάλλον στη φάση ανάγνωση από τα ανθρώπινα όντα. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα είδος ερμηνείας των δεδομένων και ένα είδος κατανόησης όχι απαραίτητα με τη γνώση. Οπότε πρέπει να κατανοήσουμε τι γίνεται με τα αισθήματα, τα συναισθήματα, τους σχετισμού το περιεχόμενο. Οπότε αυτά καμιά φορά είναι πολύ πιο χρήσιμα στις δημοσίευσεις επιστημονικές από τα απλά, τα στεγνά δεδομένα. Κάποιος λοιπόν πρέπει να διοργανώσει αυτή την πληθώρα πληροφοριών. Και όπως ξέρουμε και εμείς οι Ιταλοί με τον καφέ, ότι καλές μηχανές, αλλά ο καφές είναι εξίσου σημαντικός, όπως και η διαδικασία άλεσης και το νερό. Αν λοιπόν δώσετε πολλά χρήματα στους κατασκευαστές μηχανών, θα κάθονται εκεί στο πάλο άλτο, γιατί εκεί είναι, και θα βρουν μόνοι του. Ενώ εδώ πρέπει να δράσουμε ομαδικά. Και αυτό θα πρέπει να επιτρέπει η νομοθεσία αυτή. Ώστε να υπάρχει χρήσιμο και παληθεύσιμο περιεχόμενο. Δηλαδή να υπάρχει ο καφές, ο καφές που έχει αλεστεί, που έχει επιλεγεί και να έχουμε το, δυνατό, το καλύτερο το καφέ για το μέλλον. Και είχαμε την δήλωση ότι για τους ερευνητικούς οργανισμούς δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για το text and data mining. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχει δυνατότητα στους ερευνητές να κατεβάσουν δεδομένα μέσω αυτής της διαδικασίας. Αλλά εδώ υπάρχουν πέντε εξαιρέσεις. Και επειδή είναι ο νέος κανόνας το data mining, ε, δεν μπορούμε να απομονώσουμε κάποια εξαίρεση. Εξαίρεση είναι εξαίρεση, δεν είναι ο κανονάς. Αν λοιπόν απομονώσουμε μία εξαίρεση, απομονώνουμε και τις, ή ακυρώνουμε και τις υπόλοιπες. Οπότε, για να είναι σωστό το κείμενο των εξαιρέσεων, θα πρέπει στις πέντε εξαιρέσεις να, να δούμε ποιος εποφελείται... και ποιος είναι ο στόχος τους. Οπότε θα έλεγα να επιτρέπεται η αναπαραγωγή στα πλαίσια του text data mining. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι ένα εργαλείο το text data mining. Δεν μπορούμε να έχουμε αντιγραφή για φωτοτυπίες όπως το ίδιο εδώ αναπαραγωγή για το text data mining. Είναι πάντως δύσκολο όπως είπε και ο καθηγητής προηγουμένως να βρούμε τις σωστές συμφωνίες όπου έστω και τα προσωρινά αντίγραφα παραμένουν αντίγραφα. Πρέπει να υπάρχουν μεταβατικές, μεταβατικά αντίγραφα και θα πρέπει να δούμε την οικονομική τους αξία. Όλες οι μορφές αναπαραγωγής λοιπόν θα πρέπει να ειδωθούν προσωρινά. Αλλά στην επιστημονική ανάλυση χρειαζόμαστε περισσότερο από προσωρινά αντίγραφα. Γιατί μπορεί αυτά τα αντίγραφα ενδεχομένω να πάνε και σε λάθος χέρια ή να μην είναι χρήσιμα ή να αποθηκευτούν με τρόπο λαθασμένο και να διαγραφούν. Θα πρέπει να γνώσουμε και από μηχανέ αν αποθηκευτούν σωστά. Οπότε η πρόσβαση είναι σημαντικό στοιχείο, αλλά η εύλογη, η νόμιμη πρόσβαση είναι, σωστή, αλλά δεν πάει αρκετά μακριά. Η νόμιμη πρόσβαση μπορεί να είναι νόμιμη, αλλά μπορεί να αφορά παράνομα αποκτηθέντα δεδομένα. Αν δούμε, ας πούμε, την οδηγία για το λογισμικό και την αποθήκευση αντιγράφων με ασφάλεια, μιλά για την πρόσβαση χωρίς εξαιρέσεις. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε εξαιρέσεις που αφορούν ας πούμε τρόπους αποθήκευσης και να τη γενικεύουμε. Τώρα για το πώς ακριβώς θα διευκολύνουμε αυτό το text data mining αυτό βασίζεται στη συνεργασία. Οπότε σας παρακαλώ διαφυλάξτε τη δυνατότητα συμφωνιών με ερευνητές των πανεπιστημίων και μην κάνετε αυτές τις συμφωνίες παράνομες. Επίσης, να είναι το ναι, πρόεδρο τελειώνω, να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των νομοθεσιών. Νομίζω ότι υπάρχουν σωστά παραδείγματα σε εθνικέ νομοθεσίε όπω στη Γαλλία, στη Γερμανία, όπου υπάρχουν σωστέ και υγιεί εξαιρέσει για το text and data mining. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, κύριε Όλιβε, έξι λεπτά ε, εσείς. Πρόεδρε, εκπροσωπώ την συμμαχία copyright για την έρευνα και την εκπαίδευση. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω εκ μέρους της συμμαχίας μας. Συγχαρητήρια για το σχέδιο διηγείας. για το copyright στην εσωτερική αγορά πνευματικών δικαιωμάτων. Να τονίσω μερικά στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν. Στείλαμε το κείμενο στο Γερμανικό Υπουργείο Ανταγωνισμού για διαβούλευση. Υπάρχει μια έκθεση που μπορείτε να κατεβάσετε το διαδίκτυο. Η Συμμαχία για την Εκπαίδευση είναι μη κυβερνητική οργάνωση στη Γερμανία Ξεκίνησε το 2004 από ερευνητές, ε, ενώσεις, ε, ιδιώτες με στόχο να βελτιώσει τους νόμους για το copyright, τα πνευματικά δικαιώματα υπέρ της έρευνας και της εκπαίδευσης. Είμαστε υπέρ της πρόσβασης για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί. Θέλουμε περισσότερη αξιοπιστία, περισσότερη ισορροπία για το καλό των δημιουργών αλλά και για τους φοιτητές, για τους ερευνητές, τους επιστήμονες και ούτω καθεξής. Είναι προς το συμφέρον τη κοινωνίας η πρόσβαση. Αυτό είναι το προεξάρχον συμφέρον το οποίο υπερέχει κάθε άλλη επιχειρηματική επιδίωξης. Επιζητούμε λοιπόν το όφελος για την κοινωνία. Δύο λόγια λοιπόν για το σχέδιο και για την έκθεση. Η εξαίρεση για τους ε, εκπαιδευτικούς εκτιμώντας υπαριθμών 15. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να απολαύουν των εξής δικαιωμάτων. Τροπολογία 11. Η εκπαίδευση που παρέχεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι εκτέτως δομής και χρηματοδότησης. Πρέπει να αναγνωρίζονται ή να διαπιστεύονται ως εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία προσφέρουν εκπαίδευση. Αυτά βάσει της νομοθεσίας του κάθε κράτους μέλους. Εδώ έχουμε έναν ορισμό ο οποίος θα έπρεπε να είναι ευρύτερος. Να μην εξαρτώμεθα λοιπόν από την μορφή του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το θέμα είναι ο σκοπός, η παροχή λοιπόν εκπαίδευσης. Είμαστε υπέρ του στόχου του άρθρου 4 να βελτιωθεί η χρήση των έργων της διανοίας καθώς και οι διασυνοριακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η συμμαχία μας ενθαρρύνει την συμπερίληψη και άλλων δραστηριοτήτων για τους σκοπούς της εκπαίδευσης στην τάξη, στο πανεπιστήμιο, αλλά και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτές οι δραστηριότητες όμως πρέπει να αναφέρονται ρητός, αλλιώς δημιουργείται ασάφεια. Παλιά εκπαίδευση ονομάζαμε μόνο αυτό το οποίο γίνεται μέσα στην τάξη. Πρέπει να διευρύνουμε λοιπόν τον ορισμό. Αυτό θα αποτελέσει βελτίωση. Τροπολογία 35 την υποστηρίζουμε διότι τονίζει την σημασία της εκπαίδευσης, επιτρέπει την χρήση ψηφιακών έργων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν τονίζει τόσο πολύ το μη εμπορικός. Επίσης, άρθρο 4, πράγμα ένα αλφά και εκεί μπορούμε να βελτιώσουμε το κείμενο εκεί που λέει μέσω ασφαλούς δικτύου. Υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Αυτός ο περιορισμός μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί μέσα σε ένα κράτος μέλος, όμως απαγορεύει την διασυνοριακή ανταλλαγή. Αποτελεί λοιπόν τροχοπέδι στις διασυνοριακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το είδαμε αυτό και στη Γερμανία θα έπλετε και την λειτουργία του μόνου διαδικτυακού πανεπιστημίου στην Γερμανία. Χρειάζεται λοιπόν να επιτρέψουμε, να δώσουμε μεγαλύτερες δυνατότητες στην διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διασυνοριακά. Και να σας δώσω και μερικά νούμερα. Έχουμε 76.000 φοιτητές στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Το 10% μένει εκτός Γερμανίας, άρα ε, η διάταξη αυτή θα απαγόρευε ακριβώ την επικοινωνία με του φοιτητέ μα εκτό Γερμανία. Επίση, να μην ξεχνούμε ότι υπάρχει μια άλλη, ε, ένας άλλος περιορισμός, το ασφαλές δίκτυο. Και αυτό αντιβαίνει στις βασικές αρχές λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η μόνιμη επιτροπή για το copyright δημιουργήθηκε το 1998-1999 81 με συγχωρείτε, για να επιδιώξει εναρμόνιση μεταξύ πνευματικών συγγενικών δικαιωμάτων κλπ. Οι συζητήσεις μας πρόσφατα αφορούν τρεις ομάδες ε, δικαιούχων. Συζητούμε επίσης τις ε, εξαιρέσεις, ε, βιβλιοθήκες και αρχεία. Δεν θέλουμε η οδηγία να περιορίσει λοιπόν το δικαίωμα όλων αυτών να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω των περιορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την βελτίωση των έργων στο περιβάλλον της εκπαίδευσης είναι το άρθρο 4 παράγραφος 2. Στην Γερμανία έχουμε μια παρόμοια διάταξη, έχουμε μια εξαίρεση η οποία προήλθε από απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Το σχέδιο λοιπόν του δικού μας Υπουργείου Δικαιοσύνης λέει στο 16G η νόμιμη χρήση επιτρέπεται και ότι κάθε θέμητος περιορισμός καθιστά οποιαδήποτε σύμβαση άκυρη. Νομίζω ότι και η οδηγία πρέπει να διατυπωθεί αντίστοιχα. Είμαστε κατά των 37 και 38 των τροπολογιών. Μετά στο 6-4 ε, και εκεί πρέπει να διαγραφεί ο κανόνας διότι δεν υπηρετεί την εκπαίδευση. Θα θέλαμε επίσης να μπορούμε να χρησιμοποιούμε πολλαπλό υλικό από διαφορετικές πηγές ε, δεν είναι δυνατόν να διαπραγματεύεται κανεί με ένα σωρό διαφορετικού ε, παροχού. Άρθρο 5. Πολιστική κληρονομιά, αντίγραφα, έργων, μόνιμες συλλογέ κλπ. Πρέπει να μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο με σκοπό την διατήρηση και προστασία αυτών των έργων. Αυτό υποστηρίζεται επίσης και στα σχετικά εκτιμώντα επίσης υπέρ, του άρθρου 13, υποχρεωτική κατάθεση έργων. Στην γνωμοδότηση επίσης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς υπάρχουν ε, μερικές καλές παρατηρήσεις. Το άρθρο 5 ευτυχώς δεν προσπαθεί να προσδιορίσει τι σημαίνει πολιστική κληρονομιά, ότι υπάρχει ημερομηνία μετά την οποία τα κράτη-μέλη θα αρχίσουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια. Είμαστε υπέρ της πρόθεσης τα θεσμικά όργανα να έχουν το δικαίωμα να κάνουν αντίγραφα. Λείπει όμω ένα κανόνα σχετικά με το πώ ε, τα θεσμικά όργανα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αντίγραφα αυτά. Βιβλιοθήκε, μουσεία και αρχεία προστατεύουν βεβαίω τα έργα, αλλά προσφέρουν και πρόσβαση στο κοινό. Συνεπώ, η χρήση των αντιγράφων πρέπει να επιτρέπεται για εκπαιδευτικού σκοπού. Ιδιαίτερα όταν ε, δεν μπορούμε να επικαλυστούμε την ανάγκη διατήρηση και προστασία των έργων αυτών. Η ψηφοποίηση λοιπόν μα βοηθάει όλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα Αρνό Ρομπέρ, νομικέ υποθέσει τη ΑΣΕΤ ΛΥΒ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ομιλώ εδώ εκ μέρου τη ΑΣΕΤ. Μεγαλό ευρωπαϊκό εκδοτικό οικο στην Αγγλία, στη Γαλλία και την Ισπανία. Ο σκοπός ενός εκδότη είναι να βγάζει όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία για όσο το δυνατόν περισσότερου ανθρώπου. Αυτός είναι ο στόχος ενός εκδότη. Συγγνώμη λίγο για τον, για προκλητικό ε, τίτλο, αλλά Θέλω να συζητήσουμε λίγο το θέμα των υποχρεωτικών εξαιρέσεων στο copyright. Οι Γάλλοι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιούν αποσπάσματα από βιβλία, διηγήματα, δοκίμια κλπ. τα μετατρέπουν σε ψηφιακή μορφή χωρίς ε, να υπάρχει κανένα εμπόδιο, καμία άλλη υποχρέωση. Αυτό γίνεται ελεύθερα δηλαδή. How come? It's because... Πώς γίνεται αυτό? Τα σχολικά βιβλία, ξέρετε εμείς ε, οι εκδότες έχουμε δώσει άδειε που επιτρέπουν λοιπόν στα σχολικά βιβλία με μια μικρή αμοιβή 20 ευρώ ανά έτος Έχουν λοιπόν οι διδάσκοντες ε, απεριόριστη πρόσβαση στο υλικό με 20 ευρώ το χρόνο. Μιλούμε για χιλιάδες ε, τίτλους, η πρόσβαση είναι εύκολη. Μέσω τριών πλατφορμών ε, φιλικών προς το χρήστη μπορεί ο καθένας να κατεβάσει ό,τι θέλει. Ε, σε διάφορες συσκευές, στη συσκευή της προτιμήσεώς του ο καθένας. Τι γίνεται τώρα ε, α, όταν ένας δάσκαλος θέλει να χρησιμοποιήσει διδακτικό βιβλίο, σχολικό βιβλίο, άλλο από αυτά τα οποία έχει προβλέψει το Υπουργείο. Υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος, ο οποίος επιτρέπει στους δασκάλους να κατεβάζουν αποσπάσματα από άλλα βιβλία για τους σκοπούς της διδασκαλίας. Το κόστος αυτού είναι 11 λεπτά του ευρώ το χρόνο ανά μαθητή ανεξαρτήτως του αριθμού των αποσπασμάτων που θα κατεβάσει ο δάσκαλος. Και εδώ έχουμε λοιπόν μια εξαίρεση. Λοιπόν, δεν έχουμε εδώ περιορισμούς. Υπάρχει πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο, οπότε χρειάζεται, βάσει ατομικών ή συλλογικών αδειών. Αυτά συμπληρώνουν τις πρώτες ε, συμφωνίες που σας είπα για το, υπέρ των διδασκόντων, με την προϋπόθεση βεβαίω η χρήση να μην είναι εμπορική. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η εξαίρεση πρέπει να καλύπτει και τα σχολικά βιβλία, τα οποία φτιάχτηκαν ακριβώ για την εκπαίδευση, μια συγκεκριμένη αγορά αυτή. Δεν μπορούν όμω όλα αυτά να είναι απολύτω δωρεάν, γιατί η αγορά αυτή έχει καταστραφεί. Η εξαίρεση λοιπόν Πρέπει να είναι υπό να υπάρχουν δηλαδή οι άδειε γιατί οι άδειε έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν στην πράξη. Επίσης, η εξαίρεση δεν πρέπει να καλύπτει το σύνολο ενό έργου, γιατί δεν μιλάμε για εξαίρεση πια. Μιλάμε, εμείς θέλουμε μόνο τα αποσπάσματα να καλύπτονται. Από εκεί πέρα Πρέπει να υπάρχουν αμοιβέ για όλα αυτά, γιατί αλλιώ ένα εκδοτικό οίκο δεν βλέπω πώ θα πληρώσει υπαλλήλου, φω, νερό, τηλέφωνο κλπ. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την εκπαίδευση. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι δημιουργοί πρέπει να αμείβονται. Και όσον αφορά τι εξαιρέσει ε, που αφορούν την πολιτιστική, πολιτιστική κληρονομιά, το κράτος πρέπει να προσδιορίζει σχετικές λεπτομέρειες. Αν μια βιβλιοθήκη ή ένα μουσείο νομίζω έχει το δικαίωμα να ορίζει αυτό τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά, τότε χαθήκαμε. Πρέπει λοιπόν η αποστολή να ορίζεται πολύ συγκεκριμένα το κάθε μουσείο για παράδειγμα μπορεί να δίνει άδεια για τα δικά του έργα, αυτά τα οποία φιλοξενεί σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει και το τεκμήριο της ε, διαφύλαξης ενός πολιστικού έργου. Και τέλος, τα μη εμπορικού χαρακτήρα έργα, τα οποία δεν κυκλοφορούν πια, αυτά θα μπορούσαν να αναβιώσουν χάρη σε αυτές τις εξαιρέσεις. Βασικά εδώ δεν χρειάζεται ε, εξαίρεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, δεν χρειάζεται κανάδια. Χρειάζεται όμως να καλυφθεί το κόστο της αναπροής και τη ψηφιοποίηση αυτών των έργων που είναι πλέον εκτό κυκλοφορία. Εδώ ενδεχομένω έχουμε το θέμα των οργανισμών συλλογική διαχείρισης δικαιωμάτων και εδώ πρέπει να καλυφθεί λοιπόν ένα κόστος για να, να μπορεί να ανεβεί αυτό το περιεχόμενο σε κάποια πλατφόρμα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο τελευταίος ομιλητής για την ακρόαση και νομίζω, ε, μάλλον ευχαριστήσω τους ε, διερμηνείς για την υπομονή τους και για το χρόνο που μας χάρισαν. Ε, λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας ε, στην επόμενη ε, συνάντησή μας, μόνο αν κάποιος θέλει να κάνει μια ζωτική σημασία σε ερώτηση, τότε προφανώς μπορεί να την κάνει. Δεν υπάρχει όμω καμία τέτοιου είδου ερώτηση. Ε, Ω εκ τούτου ευχαριστώ τους ε, ομιλητές ε, που μας εμπλούτησαν με τις γνώσεις τους. Τους ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε συνάντηση των συντονιστών στις 2.30 και στις 3 κανονικά η συνεδρίασή μας. Γεια σας.